Καλημέρα σε όλους σας. Okay, when everybody has taken... Λοιπόν, αν καθίσατε όλοι, καλή σας μέρα. Αποσία της Μαρία Αρενά, η οποία έχει κολλήσει την κίνηση σε ένα λεωφορείο. Θα ήθελα να κηρύξω εγώ την έναρξη της συνεδρίασης με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχετε αντιρρήσεις, αιτήματα για αλλαγές, τροποποίησεις, όχι. Ωραία. Τότε υποθέτω ότι εγκρίνεται. Ανακοινώσεις της Προέδρου, θα σας τα διαβάσω γιατί τα έχω τώρα εδώ. Την περασμένη Παρασκευή έγιναν σημαντικές ε, διαδηλώσεις στην Αίγυπτο κατά του καθεστώτος του Πρόεδρου Ελσίση η απάντηση των αρχών ήταν βίαιη. Εκατοντάδες πολιτών, μεταξύ αυτών και ανήλικοι, συνελήφθησαν επειδή ασκούσαν το συνταγματικό τους δικαίωμα του συνέρχεστε και ε, του διαδηλώνει. Ε, Στη συνέχεια ε, τα κοινωνικά μίδια και τα blog ε, μπλοκαρίστηκαν. Καταδικάζουμε αυτή την κίνηση και καλούμε τις αρχές να αφήσουν ελεύθερους όλους τους δημοσιογράφους, διαδηλωτές, πολιτικούς αντιφρονούντες, αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικηγόρους, των οποίων δεν έχουμε νέα καθόλου. Καλούμε τις ε, Αιγυπτιακές αρχές να σέβονται το θεμητό δικαίωμα των Αιγυπτίων πολιτών να διαδηλώνουν ελεύθερα και ειρηνικά και να μην προβούν σε βία καταστολή θα εξακολουθούμε να παρακολουθούμε στενά τις ειρηνικές αυτές διαδηλώσεις παντού για την ειρήνη και τη δημοκρατία. Και ε, ασχοληθήκαμε επίσης με το Χονγκ Κόνγκ στην περασμένη συνεδρίαση και θα ανταλλάξουμε απόψεις αργότερα το απόγευμα για την Αλγερία και για το Σουδάν αρχές Οκτωβρίου. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε σχόλια, παρατηρήσεις, να κάνετε ερωτήσεις. Προχωρούμε στην έγκριση των πρακτικών. Η περασμένη συνεδρίαση ήταν στις 10 Ιουλίου. Κανονικά θα πρέπει να έχετε λάβει τα πρακτικά. Διαφωνεί κανείς. Καλώς. Εγκρίνονται και τα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής. Και προχωρούμε στην πρώτη παρουσίαση για σήμερα, που είναι ο δείκτης της Νορμανδίας που μετρά τις απειλές, την ειρήνη και την ασφάλεια. Το Παγκόσμιο Φόρουμ της ε, Νορμανδίας από τον Ιούνιο του 2018 λαμβάνει χώρα ετησίως στην πόλη Κάουν της Νορμανδίας. Συνδέεται εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια συμφωνία που έχει υπογράψει με τον Περιφερειάρχη. Κάθε χρόνο προσκαλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γίνονται μελέτες και διανέμονται. Ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου μας και οι συντάκτες των ε, εκθέσεων και των μελετών προσκαλούνται στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζας. Στα πλαίσια αυτής, αυτής της συμφωνίας συμφωνήθηκε να θεσπιστεί ο ε, δείκτης της Νορμανδίας για τις απειλές στην Παγκόσμια Στρατηγική Ασφαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μετράμε τις απειλές για την ειρήνη παγκοσμίω σε όλες τις χώρες. Επίσης, ένα εργαλείο για να εντοπίζουμε τις χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο και τις περιφέρειες που είναι πιο εύθραυστες για να βρίσκουμε τρόπο να δρούμε προληπτικά και να υποστηρίζουμε τις χώρες και τις περιφέρειες που κινδυνεύουν περισσότερο. Ο δείκτης σχεδιάστηκε και προετοιμάστηκε από το ΕΠΡΕ την Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει πληροφοριών και υποστήριξης που έδωσε το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης. Entitled Assessing... Η μελέτη που σήμερα παρουσιάζεται θα μας παρουσιάσει ε, τον ε, δίκτυ της Νορμανδίας. Ε, θα το περιγράψει και θα μας δώσει τα πρώτα αποτελέσματα. Καλωσορίζω τον κύριο Ετιέν Μπασό με μεγάλη χαρά που είναι διευθυντής στο EPRS στην Υπηρεσία Ερευνών και ήρθε να μας παρουσιάσει την εν λόγω μελέτη. Κύριε Μπαρζού. Αν θέλετε να μας πείτε περισσότερα για το εργαλείο αυτό και ποια η διαφορά του από άλλους δείκτες ειρήνης και ποια είναι τα αρχικά αποτελέσματα σε σχέση με τις σημερινές σειράξεις και πώς μπορεί να μας βοηθήσει στην κοινοβουλευτική μας δουλειά αυτός ο δείκτης και στην υποεπιτροπή μας. Σας δίνω το λόγο, παρακαλώ, κύριο Σετιέν Μπασό. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε τη δουλειά μας για το δίκτυ. Το έργο μας το ετοιμάσαμε κατά τη διάρκεια του εκλογικού διαλύματος την Άνοιξη φέτος. Και αφορά αυτά που είπατε κι εσείς, ε, ε, παρουσιάστηκε εμείς στο φόρουμ στην Κάνη της Νορμανδίας. Θα ήθελα να παρουσιάσω τους ε, συναδελφούς Ελένη Λαζάρου, Πασό και Νόζαϊ, ε, όλοι πάλι στην υπηρεσία για την πολιτική της DG Expo, της εξωτερικής πολιτικής και συνεργαστήκαμε και με ένα εξωτερικό Ινστιτούτο για την ε, ειρήνη. Γιατί θα πρέπει να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο ε, στο διεθνέ προσκήνιο για διαφορετικέ ειρηνευτικέ πρωτοβουλίε. Γιατί βασιζόμαστε ω ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στην ειρήνευση και γιατί φυσικά υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, υπάρχουν και διαφιλονικίε, όμως αυτές ε, επιλύονται εντό του θεσμικού πλαισίου και των νομικών σχέσεων που καταρτίζονται μεταξύ μας. Έχει δημιουργηθεί βεβαίως ε, μια τάση να προκύπτουν νέες ε, διανέξεις παγκοσμίω. Και όπως θα δείτε και στην εικόνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε για τη δράση της, μάλλον βλέπουμε εδώ ένα βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τις πρωτοβουλίες του στην ειρήνη, για την ειρήνη εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, το 2016, ξεκινήσαμε να θεσπίζουμε μια στρατηγική την οποία ετοιμάσαμε από την, ε, εξωτερική υπηρεσία, από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης αλλά την ενέκριναν και όλες οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Μπόρεσε να συμβάλλουν εγκαίρω. Είναι λοιπόν, θα έλεγε κανείς, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδιαιτερότητά τη είναι ότι προσπαθεί να καλύψει την περίπλοκη κατάσταση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος επικεντρωνόμενη στις απειλές. Ένα άλλο στοιχείο της δουλειάς μας έχει να κάνει με τις προσδοκίες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια σειρά από μελέτες που δεξήγαμε για το θέμα αυτό των προσδοκιών κατά τη διάρκεια του κλικού διαλύματος και μεταξύ των 15 θεμάτων που θα δείτε και στη διαφάνεια ενδεχόμενης δράσης βλέπουμε τι είναι το πιο σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες και βλέπουμε και την εξωτερική δράση να εμφανίζεται. Είναι κεντρική σημασία για τους πολίτες. Η έμφαση αυτή που δίδεται στην ε, εξωτερική δράση είναι σημαντική και για το μέλλον του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Με την ε, αύξηση της ασφάλειας και αμυνάς κεφάλαιο 5 και κεφάλαιο 6 για την ε, διεθνή συνεργασία μας. Τα βλέπετε και στις διαφάνειες δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη του δείκτη αυτή ή καθεαυτή. Αλλά είναι ένα τμήμα που έχει ετοιμάσει η Ελένη Λαζάρου για την συνολική επισκόπηση για την ειρήνη και την ασφάλεια. Ο δείκτης της Νορμανδίας μας επιτρέπει να έχουμε μια φωτογραφική απεικόνηση αναγεωγραφική περιοχή και χώρα. Ή μίλησε για την ε, σφαιρική μας στρατηγική από το 2016, γιατί το λέμε δείκτη της Νορμανδίας, διότι όπως σωστά είπατε κυρία Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο πριν από δύο χρόνια υπέγραψε μια συμφωνία εταιρική σχέση με αυτή την περιφέρεια που έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία, επειδή εκεί έγινε υποβίβαση των συμμάχων τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ε, είναι η περιοχή που έχει και την, ε, το μνημείο της ΚΑΝ με το μνημείο για την ειρήνη και ε, δέχεται χιλιάδες επισκέπτες ετησίως. Θα ρωτήσετε τώρα γιατί αυτός ο δείκτης είναι διαφορετικός. Διαφορετικός από άλλους παρόμοιους. Η ειρήνη δεν είναι απλώς απουσία διενέξεων ή συγκρούσεων. Είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο. Δεν ασχολείται ο δείκτης με το κατά πόσον υπάρχει πόλεμος ή ειρήνη σε μια χώρα ή όχι αλλά το πόσο μπορεί η ειρήνη να απειληθεί ε, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Η προστιθέμενη αξία, όπως είπατε, είναι ότι βάσει των 11 κριτηρίων της ε, σφαιρικής στρατηγικής, μερικά από αυτά είναι αρνητικά, τα 10 και ένα είναι αρνητικό, ε, θετικό συγγνώμη, η ποιότητα των δημοκρατικών διαδικασιών, αλλά βλέπετε και τις κλιματικές αλλαγές, την κυβερνοασφάλεια μεταξύ των κριτηριών, την τρομοκρατία σε διαφορετικά υποσύνολα και κλάστερ ή την οικονομική κρίση ή την ε, αστάθεια των δημοκρατικών θεσμών. Σημαντικό είναι να επισημάνουμε στη δουλειά που κάναμε ότι τα 11 κριτήρια είναι ισότιμα Όταν μελετήσαμε δείκτε ή δεδομένα που αφορούν τα διάφορα υποσύνολα τη σφαιρική στρατηγική, δεν βρήκαμε πάντα ακριβώ να αντιστοιχούν ε, τα δεδομένα με τα κριτήρια. Για παράδειγμα, στη σφαιρική στρατηγική υπάρχει και ένα κλάστερ υποσύνολο για την παραπληροφόρηση. Δεν υπήρχε κάτι σχετικό λοιπόν στα δεδομένα μας, το πήραμε ως ελευθερία του τύπου, για το οποίο έχουμε και από τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα στοιχεία για τα εγκλήματα, την εγκληματική δράση και τις εγκληματικές οργανώσεις και αυτό το εντάξαμε αλλού. Η αξιολόγηση αυτή οδηγεί σε μια χαρτογράφηση που κάναμε για τις απειλές παγκοσμίω. Βλέπετε τον χάρτη στην διαφάνεια και βλέπετε ότι οι χώρες που είναι πιο σκούρες είναι αυτές με τις σοβαρότερες απειλές κατά της ασφάλειας. και ως προς τις θέσεις των διαφορετικών χωρών. Σημαντικό είναι να πούμε ότι για κάθε δίκτυ αυτό που ισχύει είναι ότι οι αριθμοί είναι μόνο ένα σκέλος και σημαντικό είναι πάντοτε να κάνουμε και μια πιο συγκεκριμένη διεξοδική ανάλυση. Η μελέτη μας το έχει κάνει αυτό. Χώρα ανά χώρα. Πώς να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τη μελέτη. πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε το δίκτυ. Ανάλογα με τις χώρες, ανάλογα με την κάθε διάσταση. Καλημέρα σας κυρία Πρόεδρε. Ε, ή ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Αυτό που φαίνεται τώρα στο διάγραμμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πάει καλά στον κόσμο. Η πορτοκαλιά γραμμή είναι ο μέσος για τον κόσμο και το γαλάζιο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Αυτό που βλέπετε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω παρακαλώ, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ίσως λίγο χειρότερη σε τρία σημεία από άλλους για την ε, ενεργειακή ασφάλεια και την παροχή ενέργειας. Είμαστε κάτω από το μεσόρο, αλλά και για τις κλιματικές αλλαγές και την κυβερνοασφάλεια. Είμαστε πάνω από το μεσόρο. Αλλά βεβαίως και εκεί υπάρχουν κάποιες ε, αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε βάσει των όσων προκύπτουν από τα δεδομένα. Επόμενη διαφάνεια. Ο δείκτης επιτρέπει την συγκρισιμότητα και μεταξύ γεωγραφικών περιοχών είτε μεταξύ πύρων είτε μεταξύ πολιτικών οργανώσεων. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε η Λατινική Αμερική, μπορούμε να πούμε Μερκοσούρ. Για κάθε ε, περιοχή είναι δυνατόν να δούμε τη θέση τη χώρα εντό τη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη. Να, η Μακεδονία, α πούμε, και η κατάσταση της Μακεδονίας ε, σε σχέση με την υπόλοιπη Ήπειρο. Βλέπουμε που, έχει που υπάρχουν περισσότερες απειλές για τη Μακεδονία. Πιο σοβαρό από τα δεδομένα αυτά είναι να πούμε ε, ότι το σημαντικό είναι ε, η ερμηνεία των αριθμών αυτών και των δεδομένων, το κείμενο που τα εξηγεί. Βλέπετε τι έχουμε γράψει δίπλα στα αριθμητικά στοιχεία και θα δείτε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες ε, στο κείμενο της μελέτης λοιπόν. Για την περίπτωση της Ινδίας. Η Ινδία θεωρούμε ότι είναι πολύ ευπαθής σε ό,τι αφορά την ειρήνη σε πολλά σημεία και κεφάλαια. Τέλος, Και για να απαντήσω στην ερώτηση που έθεσε η πρόεδρος ε, αρχικά, τι μπορούμε να κάνουμε με τον δείκτη. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε το κοινοβουλευτικό έργο. Καταρχάς, ο δείκτης απεικονίζει τις απειλές παγκοσμίω. Αυτό ε, επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί γρήγορα και απλά. Προσφέρει πολλές πληροφορίες για την ώρα δεν είχαμε κοινή αξιολόγηση των απειλών ή κάποιο σχετικό μηχανισμό. Αλλά αν σκεφτούμε τι γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο, μπορεί να είναι και για σας ένα εργαλείο ελέγχου. Σύντομα θα έχουμε τους ακρόασει ακροάσεις για τον, είπα, το εκπρόσωπο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για άλλε διαστάσει, γειτονία, ε, ανάπτυξη, ε, ενέργεια και συνεργασία. Αυτά όταν κάποιος έχει ερώτημα για συγκεκριμένη χώρα, μπορεί να βοηθηθεί από τη μελέτη. Να δει τι γίνεται από εδώ και από εκεί, στον κόσμο, και να εντοπίσει που υπάρχουν ε, σημαντικότεροι κίνδυνοι και που πρέπει να δοθεί έμφαση στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν για μια χώρα είναι πρόβλημα η κυβερνασφάλεια, οι κλιματικές αλλαγές, φαίνεται ότι κάπως πρέπει να αναλάβουμε δράση σε αυτούς τους πολιτικούς τομείς. Επίσης για την συγκρισιμότητα. Αυτή τη ε, διάσταση θα την αναπτύξουμε περαιτέρω γιατί τα έχουμε βάλει και στο διαδίκτυο ε, με συγκέντρωση των στοιχείων σε μπάσκετ, σε καλάφια και θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να συγκρίνουμε καλύτερα μεταξύ των χωρών στο, στην παράδοση του χρόνου. Ελπίζω να το βρείτε χρήσιμο το εργαλείο θα συνεχίσουμε να το βελτιώνουμε και να το τελειοποιούμε και στο μέλλον και ελπίζουμε ότι θα μπορούμε να κάνουμε και άλλες συγκρίσεις, ακόμα καλύτερες, βελτιώνοντας το περιεχόμενο της μελέτης, όπως είπα για την κυβερνοασφάλεια, και για τα διασυνοριακά εγκλήματα θα πρέπει να δούμε τι δεδομένα μπορούμε να συγκεντρώνουμε και στο μέλλον. Έχει γίνει πολύ ποιοτική δουλειά με συνεργασία όλων των συναδέλφων από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου ε, και ευχαρίστως να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Όλοι έχουμε μπροστά μας την μελέτη που μας απεστάλλει ηλεκτρονικός θα μπορούμε να τα μελετήσουμε. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ξεκινήσω με την Ιζαμπέλ Βίσλερ και μετά η κυρία Ντουσάντος. Bonjour, Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μπασό και όλη την ομάδα του για όλη αυτή την εργασία που έκαναν που σίγουρα απέτησε πολλή ενέργεια, πολλή προσπάθεια. Σε λίγα λεπτά καταφέρατε να μας παρουσιάσετε ένα τεράστιο έργο. Το πρώτο μου ερώτημα είναι το ακόλουθο. Προβλέπετε, μάλλον, πώς θα γίνεται η επικαιροποίηση του δίκτυα αυτού, γιατί αν κατάλαβα καλά έχουμε μία απεικόνηση αυτή τη στιγμή, μία φωτογραφική απεικόνηση της τρέχουσας κατάστασης, πώς θα ενημερώνεται αν θέλετε η εικόνα αυτή, πώς θα την επικαιροποιούμε γιατί μόνο αυτό θα μας επιτρέψει τελικά να κάνουμε πραγματικές συγκρίσεις ανάμεσα στις διάφορες χώρες και να βλέπουμε και τη σχετική εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης. Πέρα από αυτό, μου έκανε εντύπωση κάτι το οποίο αναφέρατε, κάτι το οποίο μας ανησυχεί όλους ιδιαιτέρως, το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ως προς αυτό είπατε ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα, ότι εσείς χρειάστηκε να αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα διότι σε κάθε περίπτωση δεν καταφέρατε να σημειώσετε την πρόοδο που θέλατε στον τομέα αυτό. Επομένως, σας ρωτώ τι παραπάνω πρέπει να κάνουμε, προκειμένου να έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με τον τομέα αυτό. Να αφήσω επίσης το λόγο και στους υπόλοιπους συναδέλφους για να κάνουν και αυτοί κάποιες ερωτήσεις και περιμένω και την απάντησή σας κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ιζαμπέλ Σάντος, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πρωτογαλλικά. Επομένω, φορέστε τα ακουστικά σας, παρακαλώ. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπασό και την ομάδα του για την ε, πολύ καλή δουλειά που μας παρουσίασαν εδώ και που είναι πραγματικά πολύ καλή αφετηρία και θεμέλιο για την αξιολόγηση της κατάστασης στον κόσμο σε ό,τι αφορά την, τις απειλές κατά της ειρήνης και της ασφάλειας. Πολύ καλή, καλός τρόπος για να υποστηρίξουμε και να θεμελιώσουμε την πολιτική μας δράση όπως τη σχεδιάζουμε και όπως την ε, χαράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωταγωνιστή στην παγκόσμια ασφάλεια και την εγγύηση της ειρήνης. Η μελέτη αυτή προφανώς θα αλλάξει στο μέλλον και όταν την κοιτάζω προσεκτικά και επειδή υπάρχει και μια διάσταση κοινωνιολογική σε όλα αυτά, εδώ βλέπω να γυρώνται απευθείας κάποια ερωτήματα. Ο κύριο Μπασό δεν το εμβάθυνε το θέμα για την παραπληροφόρηση. Το θίξατε, αλλά δεν εμβαθύναμε. Η παραπληροφόρηση είναι σταθερά μια απειλή κατά τη ειρήνης και της ασφάλεια. Είναι μια απειλή κατά της εμπιστο... του κλίματος εμπιστοσύνη εντό των χωρών. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε μελλοντικά τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει και τι δράση να αναλυθεί για τα θέματα της παραπληροφόρησης. Θέματα που όλο ένα και περισσότερο απασχολούν. Και σε συνδυασμό με την ερώτηση που έκανε η συνάδελφος, η Ζαμπέλημα, ήθελα να μου πείτε για την κυβερνοασφάλεια Ποιε πραγματικά δυσκολίε είχατε στο να συγκεντρώσετε στοιχεία για το θέμα αυτό, Έλλειψη δεδομένων, έλλειψη συνεργασία από τους διάφορους φορείς που χειρίζονται τα δεδομένα, δεν σας ε, παρήχαν ε, πληροφορίες. Πού είναι ακριβώς η μεγαλύτερη δυσκολία σε αυτή τη διάσταση. Και ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα για το διασυνοριακό έγκλημα. Ξέρουμε ότι οι απειλές ε, δεν γνωρίζουν σύνορα και τα υπερπηδούν διαρκώς όλο και περισσότερο. Στη μια ή στην άλλη περιοχή σημείο της επικρατειάς μας. Μπορείτε να μας πείτε δύο πράγματα και γι' αυτό. Γιατί μου φαίνεται πραγματικά κέρια σημασίας για το πώς έχετε κι εσείς ε, καταρτήσει την ε, όλη σας προσέγγιση για την αξιολόγηση της περιοχής μας και του υπόλοιπου κόσμου ως προς την ασφάλεια και την ειρήνη. Ε, Ευχαριστούμε. Η Ρεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ήθελα να συμφωνήσω με τα σχόλια των προλησάντων. Όντω, η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχετε κάνει μια τεράστια εργασία για την κατάρτισή της. Έχω μια ερώτηση όσον αφορά την εξέλιξη των κινδύνων και των απειλών σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώ και έχουμε εξέλιξη των απειλών και των κινδύνων σε καθημερινή, θα έλεγα, βάση. Με βάση τα κριτήρια λοιπόν τα χρησιμοποιείτε, πώ καταφέρνετε να επικυρωποιείτε την έκθεση αυτή και με τι συχνότητα κάνετε αυτή την επικυροποίηση και πώ μπορούμε, για παράδειγμα, να διασφαλίσουμε ότι ε, μια σημαντική αλλαγή στον εκτιμόμενο κίνδυνο μπορεί πραγματικά να φτάσει σε εμά, να λάβουμε γνώση για αυτήν το στομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κατρίν Χάβιτ. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή. Και οφείλω να πω βέβαια ότι διατηρώ μια σκεπτική στάση ακόμα. σε σχέση με την καταλληλότητα της έκθεσης αυτής και του όλου αυτού εγχειρήματο το να κάνουμε μία τόσο μεγάλη και σημαντική από ποσοτική πλευρά ανάλυση, χρησιμοποιώντα τόσα πολλά διαφορετικά δεδομένα και πολλέ διαφορετικέ στατιστικέ μεθόδου. Να επικεντρωθώ απλώ σε κάποια ζητήματα. Αν για παράδειγμα αυτό ήταν ε, μια διδακτορική μελέτη που μου παρουσιαζόταν, θα ζητούσα πάλι από το φοιτητή να αρχίσει πάλι μια ολόκληρη έρευνα για να δει πραγματικά ποια είναι τα κριτήρια αυτά τα οποία χρησιμοποιεί και αν ορισμένα κριτήρια τελικά μπορεί να στρεβλώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Μήπως θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποια πιο αντικειμενικά κριτήρια, για παράδειγμα. Είναι σαφές αυτή τη στιγμή ότι όντως ασχολούμεθα με τις χώρες αυτές οι οποίες ε, τελούν υπό απειλή στις απειλές αυτές καθεαυτές. Και αν ασχολούμεθα με τις απειλές, ασχολούμεθα με τους υπέτειους για τις ε, απειλές αυτές ή για τους ανθρώπους εκείνους ή τις χώρες εκείνες οι οποίες τελούν υπό απειλή. Για παράδειγμα, βλέπω στον κατάλογό σας ε, την Παλαιστίνη στην θέση 56 για παράδειγμα. Βλέπω και τη Βραζιλία εν συνεχεία στην θέση 45 του καταλόγου σας πώς μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο και πώς μπορεί ο κατάλογος αυτός να είναι εύστοχος και κατάλληλος για μας και να αποτελεί βάση εργασίας τη στιγμή που έχουμε αυτή την βαθμολόγηση, αν θέλετε, των κρατών σε σχέση με τις απειλές και δούμε τους βασικούς εισαγωγείς όπλων επίσης. Μήπως θα έπρεπε επίσης να επικεντρωθούμε κυρίως στα συμβατικά όπλα και όχι αναγκαστικά στα όπλα μαζικής καταστροφής. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, θεωρείτε ότι η Σεδική Αραβία δεν ανήκει στις χώρες εκείνες οι οποίες απειλούν την παγκόσμια ειρήνη. Νομίζω ότι όντω η προσέγγιση σας είναι προβληματική σε κάποια σημεία και τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιείτε για να καταρτήσετε τον κατάλογο αυτό ουσιαστικά είναι κριτήρια τα οποία αναμειγνύουν τόσο τις απειλές όσο και τους απειλούμενους. Από την απτική τώρα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομίζω ότι τα όσα λέτε για την ελευθερία του τύπου, το σχετικό κριτήριο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο για την αποτίμηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια χώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι χρησιμοποιούνται κάποια κριτήρια και έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι που εγείρουν κάποιες ανησυχίες. Ενδεχομένως θα μπορούσατε να έχετε χρησιμοποιήσει τον χρόνο που αφιερώσατε ε, στο να κάνετε μια πιο ποιοτική έρευνα και να αναλάβετε μια πιο ποιοτική δράση που θα ήταν πιο χρήσιμη τελικά και για μας. Πίτερ Βαντάλεν, παρακαλώ. Ε, θα μιλήσω Ολλανδικά, κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρία Πρόεδρε, και εγώ δεν Είμαι ικανοποιημένο πάρα πολύ από την έκθεση αυτή για διάφορου λόγου. Πρώτον, λείπει ένα πολύ σημαντικό κριτήριο που είναι το κριτήριο τη ελευθερία τη ε, θρησκεία και τη σκεφτική λατρεία. Στην σελίδα 6, α πούμε, θα ήταν τελείω διαφορετικό ο κατάλογο αν είχε συμπεριληφθεί αυτό το κριτήριο τη θρησκευτική ελευθερία. Και ε, πραγματικά είναι πολύ μονομερής και χρωματισμένη αυτή η λίστα, κατά την άποψή μου ας πούμε, η Ινδονησία είναι στη θέση 44, στην πράσινη υποτίθεται ζώνη και δεν συνιστά απειλή. Αν κοιτάξετε όμως το θέμα αυτό της θρησκείας, τότε κατρακυλάει στον πάτο, ε, στα, στην κόκκινη ζώνη η, η Ινδονησία. Η είναι στη θέση 10 οικονομικά και χρηματοοικονομικά είναι εξαιρετικά ασταθής ε, ε, επίσης ελέγχεται και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Βενεζουέλα είναι στη θέση 96, ε, στην κίτρινη ζώνη. Ο άνθρωπος είναι δικτάτορας, έχει καταστρέψει τη χώρα του, είναι καθημερινός ο πόλεμος εκεί, τους ρίχνει στη φυλακή. Στον πάτο πρέπει να είναι η Βενεζουέλα, το ίδιο ισχύει για την Κίνα. Ε, κυνηγάει τους ε, τους βάζει στη φυλακή, κλείνει διάφορες εκκλησίες. Δεν υπάρχει ελευθερία ε, της ε, θρησκευτικής λατρείας. Και αυτή είναι στην κίτρινη ζώνη. Δεν μπορούν να ισχύουν αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ μονομερής, μεροληπτική έκθεση, λαμβάνω γνώση, αλλά κρατάω και μικρό καλάθι. Ε, πολύ μονομερής προσέγγιση της πραγματικότητας, κατά την απόψή μου και ε, προκατηλημένη. Ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε, αλλά δεν μπορώ να την υιοθετήσω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαχιανή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπασό για την ε, παρουσίαση της έκθεσής του. Ε, γνωρίζω ότι είναι δύσκολη η έκθεση και όταν δει τον κατάλογο κανείς, πάντα όλοι θα έχουμε κάποιες ε, παρατηρήσεις. Επιτρέψτε μου για μερικές χώρες. Βοσνία, Ζεγοβίνη δεν γίνεται αναφορά στις τζιχατιστικές ομάδες, μα είναι πολλοί οι ξένοι μαχητές από τη Βοσνία που βρίσκουμε στη Συρία μεταξύ άλλων. Για την Κίνα η έκθεση μιλάει για ιδιαίτερη απειλή που συνιστούν ε, οι Ουιγούροι, οι αποσχιστές για την Ινδία, εντάσεις με το Πακιστάν και ιδιαίτερα ε, η διένεξη στο Κασμίρ γέννησε ε, μια σειρά Ισλαμιστικές ομάδες που δρούν από την Πακιστανική επικράτεια. Για τη Βόρεια Μακεδονία λέει ότι η Ελλάδα σταμάτησε το βέτο ε, για το αν θα μπει στο ΝΑΤΟ η Βόρεια Μακεδονία. Αυτό είναι παράγον ασφάλειας η ένταξη στο ΝΑΤΟ ή μήπως θα υπάρξει νέο χάσμα στην Ευρώπη. Για τη Ρωσία τονίζει η έκθεση τη σημασία των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αντίπεινα ε, της Ρωσίας ε, για, ε, στη Ρωσία μάλλον για την απαγόρευση εισαγωγών γεωργικών προϊόντων, εγώ νομίζω ότι θα βοηθήσει για την ασφάλεια και την ειρήνη στην Ευρώπη άρση των κυρώσεων. Για τη Συρία, τι αριθμητικά στοιχεία έχετε και ποιος σας τα δίνει. Είναι το περίφημο παρατηρητήριο του Λονδίνου ή έχετε και άλλες πηγές, γιατί είναι πάντα αφιλεγόμενα. 63% λέει των θανάτων οφείλονται στο Ισλαμικό κράτος. Ναι, αν προσθεθούν και άλλες ομάδες Αλ-Κάιντα, Αλ-Νουσρά, αυξάνεται το ποσοστό αυτό. Ε, και με εκπλήσει η φράση που λέτε ότι ο πόλεμος και ιδιαίτερη ε, αστάθεια ε, του καθεστώτος Ασάντ κατέστρεψαν τη Συρία. Ε, δεν έχουν βάλει το λιθαράκι τους και τίποτα τρομοκράτες εκεί πέρα. Το λιθαράκι το λέω γκόλιθος, είναι ηρωνικά. Ε, και το ΠΚΚ ε, είναι η πιο... Ε, θανατηφόρα ε, ε, ομάδα ε, τρομοκρατική στην Ευρώπη εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο ζητούν κάποιοι να βγει από τη λίστα. Για την Ουκρανία, τι γίνεται με τα πολλά θύματα στην κοιλάδα του Ντόν, στον Ντόν Πας που είναι ρωσόφων. Από τις 25 χώρες που αναφέρεται, οι μισές ε, απειλούνται από ένα μεγάλο κίνδυνο που είναι ο, ο ε, ριζοσπαστικός Ισλαμισμός. Αυτό το κριτήριο της θρησκείας στο μέλλον καλό θα ήταν το συμπεριλάβετε. Και να ρωτήσω και κάτι έτσι εμπαρόδο για να τελειώσω. Πόσο κάνει η μελέτη αυτή, πόσο μας στοιχίζει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδώσω το λόγο στον Ετιέν για να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ένα δεκάλεπτο το πολύ. Το πολύ. <coughs> Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε σας, ευχαριστώ πολύ κύριε, και κύριοι βουλευτές. Ωραία, θα προσπαθήσω να απαντήσω ομαδικά για την κυβερνοασφάλεια. Η πηγή που χρησιμοποιήσαμε είναι ο Οργανισμός Διεθνών Επικοινωνίων από τη Γενέβη που έχει αριθμητικά στοιχεία για, με δεδομένα, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια κατηγοριοποίηση αναχώρα για την ε, αντίσταση, την ανθεκτικότητα κατά της παραπληροφόρησης. Για την ανθεκτικότητα αυτή δεν έχουμε κάποιον δείκτη προς το παρόν. Ε, και το είπαμε και ειλικρινώς ως προς αυτό. Χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα των ε, δημοσιογράφων χωρίς σύνορα για την ελευθεροτυπία. Δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο δείκτης. Όμως μας απασχολεί όπως και για την κυβερνοσφάλεια για να επικυροποιήσουμε τη συλλογή των δεδομένων. Πολλά ερωτήματα αφορούσαν την ε, επικαιροποίηση, το πόσο είναι επίκαιρα τα δεδομένα της μελέτης. Θέλουμε να υπάρχει η επικαιροποίηση και να μπορούμε να συγκρίνουμε από τη μια χρονιά στην άλλη, ώστε να μπορούμε να, είμαστε, να θεωρήσουμε ότι είμαστε και ε, πολύ ενεργοί εδώ. Μιλήσατε για τους αριθμούς. Όταν ξεκινά κανείς μια τέτοιου είδους μελέτη, προφανώς βρίσκεται και εκτεθειμένος διότι πρέπει να βάλει σε, μια, σε κατηγορίες και σε μια ιεραρχία τις χώρες και να βαθμολογήσει ένα ως δέκα τις απειλές της, κατά της ειρήνης. Πρέπει όμως να κοιτάξει προσεκτικά και αναλύσεις ποσοτικές. Γι' αυτό για 20 χώρες έχουμε ετοιμάσει και επιμέρους δελτία ώστε να εξηγήσουμε κι άλλες ε, λεπτομέρειες με αριθμητικά στοιχεία καλύτερα αναλυμένα. Με την ε, ομάδα κριτηρίων, αυτό το καλάθι κριτηρίων θέλουμε να δημιουργήσουμε είπαμε ότι και αντικειμενικά και θεσμικά έχει αναγνωριστεί ότι η σφαιρική στρατηγική του 2016 επιβάλλει κάποια κριτήρια. Έτσι ε, επιλέξαμε τα 11 κριτήρια. Είναι αυτά τη σφαιρική στρατηγική, του Global Strategy. Ε, τότε είχε εγκριθεί και από το Ευρωκοινοβούλιο η στρατηγική αυτή και από το σύνολο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Αυτό απετέλεσε τη βάση. Είναι προφανές ότι κάποια σημεία σε αυτή την παγκόσμια στρατηγική είναι πιο σημαντικά από άλλα. Αναφέρατε την ανεξιθρησκεία, ας πούμε, την ελευθερία της ε, θρησκευτικής λατρείας, ε, που δεν είναι απευθείας απειλή, αλλά θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα παράγοντα. Υποθέτω και σε λίγους μήνες θα έχουμε κάποιον άλλον ε, το εκπρόσωπο, μπορεί να μεταρρυθμιστεί η παγκόσμια στρατηγική. Φέτο του χρόνου θα χρειαστεί επικαιροποίηση όταν γίνει και η σχετική αλλαγή. Τώρα για την ερώτηση η ερώτηση για το κατά πόσον πρόκειται για απειλές κατά των χωρών που δέχονται αυτές απειλές. Ναι, είναι απειλές εις βάρος των χωρών. Και αυτό το ορίζει η παγκόσμια στρατηγική. Ε, χώρες κατά με απειλές που τις βαρύνουν. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές. Και τέλος για τους δείκτες μπορεί να μεταβληθούν. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θέλουν να προσθέσουν κάτι για τις αναλύσεις των επιμέρους χωρών, τα δελτία των χωρών. Ελένη. Ευχαριστώ για αυτές τις ερωτήσεις. Πάρα πολύ χρήσιμες για μας, ε, διότι θέλουμε και τη δική σας αντίδραση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τη μελέτη. Είναι πιλωτικός ο χαρακτήρας του, της μελέτης. Μαζί με την περιφέρεια της Νορμανδίας αποφασίσαμε να ε, συντάξουμε αυτή την έκθεση ω μια πρώτη δοκιμή. Γι' αυτό μα ενδιαφέρει πολύ η άποψη των βουλευτών. Τώρα, μέρο των δικτών, όπω εξήγησε και ο διευθυντή μου, δεν ήταν δική μα επιλογή. Η παγκόσμια στατικική, η προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει κάποια πράγματα. Πρέπει να ελέγξουμε και να ξεκριβώσουμε το τι συμβαίνει βάσει των όσων η ΑΕΔ έχει ορίσει ω παγκόσμιε απειλέ κατά τη ειρήνη και επί των οποίων έχει αποφασίσει να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αντιδράσει σα στην έκθεση αυτή δείχνουν ότι για του περισσότερου δείκτε δηλαδή δείχνουν ότι το θέμα είναι πώς να, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί. Το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να πει στην επατή εκπρόσωπο ποιε είναι οι απειλέ που θεωρούν ότι είναι σοβαρέ. Αν θεωρείτε ότι ότι κάτι λείπει εδώ, το, ο τρόπο για να προσθεθεί είναι να συζητήσετε με την ΕΕΔ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πείτε θεωρούμε ότι εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό ή αυτό θα πρέπει να θεωρούμε ω απειλή. Τώρα για τι ανησυχίε σα και για για να είμαστε μεθοδολογικά σωστοί, βασιστήκαμε σε δείκτες, τους οποίους συμπεριλάβαμε σε ένα καλάθι, για να το πω έτσι, το οποίο αναφέρεται και στο έγγραφο. Είπατε ε, για την ε, ακαδημαϊκή διάσταση του θέματος ε, κάποια από εσά. Μπορείτε να έχετε διαφορετικέ κατηγοριοποιήσει των χωρών με διαφορετικού βαθμού, αλλά πρέπει κανεί να καταλάβει και τι σημαίνει εδώ θέση τη κάθε χώρα στον κατάλογο. Το να είναι κανεί ψηλά ή χαμηλά στον κατάλογο έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο καλάθι δικτών. Δηλαδή, κάποιε χώρε μπορεί να μην είναι δημοκρατικά άψογε ή να έχουν προβλήματα απολυταρχικού καθεστώτο, όμω με αυτέ τι 11 μεταβλητέ ε, πρέπει να τις ταξονομήσουμε έτσι αναλόγως. Μπορεί να πηγαίνουν καλά στα θέματα του κλίματος, είναι ενεργειακά ασφαλείς. Αυτό δεν έχει να κάνει με την πολιτική του ίσως, αλλά με τη γεωγραφική του θέση. Οπότε ευχαρίστως, αν θέλετε, ως ερευνητές να μιλήσουμε ε, κατά μόνας με τον καθένα από εσά που έχει κάποιο πρόβλημα, να εξηγήσουμε γιατί μια χώρα κατηγοριοποιήθηκε με τον ένα τον άλλο τρόπο και έχουμε και όλο το ιστορικό της ερευνά μα που εξηγεί γιατί κάθε χώρα μπήκε σε μια συγκεκριμένη θέση στον κατάλογο. Βεβαίως, τις μεταβλητέ αυτές τις μελετούμε και σίγουρα είναι το αδύναμο σημείο τη έρευνά μα, γιατί όπω είπε και ο διευθυντή μας, για συγκεκριμένε μεταβλητέ, για συγκεκριμένου δείκτες δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία να παρέχονται ε, και τα οποία να θεωρούμε αξιόπιστα και να τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι πληροφορίες που κανεί ω σήμερα δεν τα έχει μετρήσει. Είναι νέες απειλέ, οπότε... Ε, Υπάρχει προσπάθεια να αρχίσουν να συγκεντρώνονται δεδομένα για αυτά, αλλά προ στιγμή δεν έχουμε κάτι το αξιόπιστο και το ανεξόρτητο που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για τη δουλειά του Κοινοβουλίου. Φίλιπ, θε να προσθέσει κάτι. Ναι, ευχαριστώ. Καταρχά να πω ότι στο σύνολο αυτή τη δουλειά αντιμετωπίσαμε δυσκολίε, κυρίω μεθοδολογία και σωστά υπογραμμίστηκε το θέμα των διασυνοριακών εγκλημάτων ψάξαμε, κοίταξαμε τα στοιχεία της Interpol και άλλων οργανισμών, σήμερα δεν υπάρχει μέτρηση των διασυνοριακών εγκλημάτων στα εκατοντάδες σύνορα που υπάρχουν, στις εκατοντάδες χώρες του κόσμου. Είναι μια εγγενής δυσκολία. Και βεβαίως, ως ερευνητές, αυτό που θα θέλαμε είναι να βρούμε τα ε, πιο αντιπροσωπευτικά στοιχεία. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στην επικαιροποίηση με κάποια από τα δεδομένα, την παραπληροφόρηση, τα διασυνορικά εγκλήματα είναι σημαντικό. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι για την κατηγοριοποίηση των χωρών, την ιεράρχηση. Δεν νομίζω ότι να επικεντρωθείτε σε αυτό, αλλά το κατά πόσον μπορούμε να έχουμε γρήγορα δεδομένα. Εσείς ως βουλευτές θα πρέπει να μπορείτε να δείτε ποιοτικά τις διαστάσεις ε, τις πιο ευάλωτες κάθε χώρα. Να πάρω δύο χώρες με την ίδια βαθμολόγηση. 19 και 2. Κώστα Ρίκα και Γεωργία. Εάν δούμε πραγματικά το προφίλ των δύο αυτών χωρών, έχουν τα δύναμα σημεία τους και τα ε, δυνατά, ε, τα πλεονεκτήματά τους. Αλλά καταλήγουν στην ίδια θέση, στην ίδια βαθμολογία στον κατάλογο. Θα πρέπει όμω κανεί να κάτσει μετά να αξιολογήσει προσεκτικά με το καθένα από τα κριτήρια τι γίνεται στον κάθε χώρα. Και όπω το είπε και η Ελένη και ο κύριο Μπασό, όλα τα δεδομένα θέλουμε να είναι στο δυνατόν διαφανέστερα και χρήσιμα. Να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε γρήγορα. Αυτό γιατί και η AI έχει το δικό τη εργαλείο ανάλυση. Αλλά τα δεδομένα αυτά δεν είναι προσβάσιμα στο κοινό. Εμεί αυτό θέλαμε να κάνουμε, να δημοσιώσουμε στα τώρα για την ελευθερία τη θρησκευτική έκφραση. Δεν ορίζεται πουθενά στην παγκόσμια στρατηγική, όμω είναι κάτι που εμεί ε, στι ερευνητικέ μα υπηρεσίε ε, το Έχουμε ήδη μελετήσει. Πριν από ένα χρόνο ετοιμάσαμε μια μελέτη και μόλι επικαιροποιηθεί θα σα το αποστείλουμε. Θρησκεία στην εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι όταν μιλάτε για θρησκευτική ελευθερία αναφέρεστε σε ελευθερία διαφορετικών πεπιθήσεων, έτσι δεν είναι, με ένα, μια προσέγγιση πιο σφαιρική, πιο γενική. Ας ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, που ανέφεραν πολύ συχνά οι συντάκτε τη έκθεση αυτή ω βασικό του εταίρο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ρενένε Φανένσεν ονομάζομαι και είμαι επικεφαλή του τμήματο εκείνου που ονομάζεται Πρόληψη Συγκρούσεων και υποστήριξη στην διαμεσολάβηση στα πλαίσια πάντα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και όντω επικεντρωνόμαστε τόσο στη μεσολάβηση, τη διαιτησία, όσο και στην πρόληψη των συγκρούσεων. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τον δείκτη τη Νορμανδία, προφανώ το χαιρετίζουμε και χαιρετίζουμε οποιαδήποτε απόπειρα γίνεται που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πρόληψη των συγκρούσεων και των διενέξεων. Σαφώ χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά που θα μα επιτρέψουν να καταλάβουμε πώ μπορούμε να αποτιμήσουμε τον κίνδυνο εμφάνιση μια βίαιη σύγκρουση Ποιοι είναι δηλαδή οι δείκτε αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν πραγματικά να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς προκύπτουν οι συγκρούσεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να συνδέσουμε όλη αυτή την ανάλυση με τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε μεγαλύτερη λεπτομέρεια πώ βαθμολογούνται οι διάφορε χώρε. Προφανώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση προσεγγίζει διαφορετικά τι συγκρούσει. Έχουμε ένα σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση που χρησιμοποιεί 25 δείκτε, οι οποίοι επικυρωποιούνται συνεχώ και βασίζονται σε συστηματικέ έρευνε, τι οποίε διεξάγουμε εμεί. Και προσπαθούμε επίση να εξετάσουμε και πτυχέ όπω το περιβάλλον. Πώ περιβαλλοντικοί παράγοντε και περιβαλλοντικέ μεταβλητέ μπορούν να οδηγήσουν σε απειλέ που στη συνέχεια θα οδηγήσουν σε συγκρούσει. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά να μπορούμε να εντοπίζουμε τις συγκρούσεις και να καταλαβαίνουμε και τα βαθύτερα αιτιά τους. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες και την ενέργειά μας σε συγκεκριμένους τομείς αν πραγματικά θέλουμε να ευοδοθεί η όλη προσπάθεια πρόληψης των συγκρούσεων. Εκτιμούμε λοιπόν όλους ιδιαίτερο συνεργασία που έχει γίνει. Όπως υπόθηκε από τους προελίσσαντες, η ανάλυση είναι πάρα πολύ σημαντική. Το τονίζω και εγώ αυτό. Ένα πράγμα είναι τα δεδομένα, προφανώ θα πρέπει να υπάρχουν δεδομένα. Εν συνεχεία, βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει μια λεπτομερή ανάλυση τη κάθε χώρα. Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, συνεργαστήκαμε και θέλουμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον με την Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να συμβάλλουμε και εμεί περισσότερο στην όλη αυτή εργασία. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτή τη συζήτηση αυτή, γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει λίγο. Πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη μελίσια διάταξη. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι παρουσιάσει που κάνατε και καταλάβαμε ότι είστε στη διάθεσή μα προκειμένου να βαθύνουμε περισσότερο σε κάθε χώρα ξεχωριστά στα πλαίσια της ποιοτική αυτής προσέγγισης η οποία σαφώς είναι σημαντικότατη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όλη εργασία σας. Περνάμε στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με την Frontline Defenders Ξέρετε σήμερα ότι μειώνεται όλο και περισσότερο ζωτικό χώρο κοινωνία των πολιτών και υπάρχουν σαφή προβλήματα όσον αφορά του υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα πρέπει ήδη από σήμερα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το ζήτημα αυτό με συγκεκριμένου καλεσμένου οι οποίοι θα μπορέσουν να μα δώσουν μια πραγματική εικόνα τη κατάσταση επιτόπου όσον αφορά τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλους εκείνους από την κοινότητα των πολιτών οι οποίοι προσπαθούν να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας καλώ να έρθετε εδώ πέρα και να δώσω καταρχάς το λόγο στην Έμα Ατσίλη, η οποία είναι υπεύθυνη του Ευρωπαϊκού Γραφείου της οργάνωσης Frontline Defenders. Θα μας γίνει μια πρώτη παρουσίαση λοιπόν από την καλεσμένη μας και στη συνέχεια θα έχουμε και δύο μάρτυρες, δύο μαρτυρίες από δύο επιτόπου ακτιβιστές οι οποίοι διαστροποιούνται στο Μεξικό, τον Παύλο Λόμπε Σαλβάρες, ο οποίος είναι ένας ακτιβιστής, ο οποίος εδώ και 9 χρόνια βρίσκεται στη φυλακή εξαιτία της όλης δραστηριοποίησής του στην πολιτεία Οξάκα του Μεξικού, κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους. Να δώσω όμως καταρχάς το λόγο στην κυρία Έμα Ακύλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω στα γαλλικά και έπειτα θα κάνω την παρουσίασή μου στα αγγλικά. Ειλικρινά λοιπόν να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ε, μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε μια γενική συζήτηση όσον αφορά την κατάσταση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άνθρωποι ιδιαίτερα θαραλέοι, έχουμε και δύο καλεσμένους εδώ πέρα, άνθρωποι οι οποίοι με ιδιαίτερο θάρρος, ιδιαίτερη αποφασιστικότητα και κινδυνεύοντας πάρα πολλά πράγματα καταφέρνουν να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχουμε πάρα πολλού οι οποίοι υπερασπίζονται του υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Γιολάντα ήρθε από το μακρινό Μεξικό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει περισσότερο στο κέντρο τη δράση του του υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του προφανώ. Ε, σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σα, κυρία Πρόεδρε να μα καλέσετε σήμερα εδώ. Θα συνεχίσω τώρα την παρουσίασή μου στα αγγλικά. Έχουμε μία παγκόσμια ανάλυση, θα μπορούσα να σας δώσω και περισσότερα αντίγραφα της έκθεσης μας αυτής, η οποία περιγράφει την κατάσταση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Δυστυχώ όμω τα νέα δεν είναι ιδιαίτερα χαρμόσυνα όσον αφορά τι αναδυόμενε τάσει για του περασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πλέον σαφέ ότι ε, απειλούνται όλο και περισσότερο οι περασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι καταπατώνται όλο και περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2018 εμείς ε, αναφέραμε την δολοφονία 321 υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια των εκθέσεών μας. Πρόκειται για δεδομένα τα οποία είναι ακόμα μερικά, δεν έχουμε πλήρη εικόνα των δολοφονιών αυτών. Ενδεχομένω θα ήταν σημαντικό να καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε και περαιτέρω έρευνες για περαιτέρω δείκτες. Όσον αφορά τις δολοφονίες, έχουμε, αν θέλετε, τις ίδιες πάντα χώρες που εμφανίζονται στην έρευνά μας, η Κολομβία, το Μεξικό, Φιλιππίνες και Βραζιλία. Πρόκειται για τις χώρες εκείνες που έχουμε τις περισσότερες δολοφονίες, αλλά και τα περισσότερα φαινόμενα καταστολής που έχουν να κάνουν κυρίως με τα δικαιώματα στην έγκυη ιδιοκτησία, στην, στα περιβαλλοντικά δικαιώματα, στα δικαιώματα των αυτόχθονων ανθρώπων. Ένα 77% των όσων θανατώθηκαν εργάζονταν στους τομείς αυτούς και έχουμε και μια αύξηση σε σχέση με το 67% που είχαμε το 2017. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι στι περιοχές αυτές κινδυνεύουν τρει φορές περισσότερο να χάσουν τη ζωή του, σε σχέση με περασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλες περιοχές του κόσμου ή σε άλλου τομείς. Χρειαζόμαστε λοιπόν εμείς την απαραίτητη χρηματοδότηση και την υποστήριξη θεσμική και από τις κυβερνήσεις προκειμένου να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα βίας κατά των περασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν υποτίθεται ότι παρεμποδίζουν πολύ σημαντικά έργα ή όταν προσπαθούν να προασπίσουν τα δικαιώματα χρήσης γης συγκεκριμένων αυτόχθονων ανθρώπων. Η Γιολάντα που είναι εδώ πέρα δίπλα μα δραστηριοποιείται ακριβώ στον τομέα αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερο τους ανθρώπους αυτούς ως συμμάχους μας για την προστασία του περιβάλλοντο και για το μετριασμό ή την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Οι δολοφονίες αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί και το, σε ένα ποσοστό 90% των δολοφονιών αυτών είχαν προηγηθεί συστηματικές απειλές εναντίον των περασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυστυχώς όταν οι άνθρωποι αυτοί πήγαν σε αρμόδιες αρχές για να καταγγείλουν τις απειλές αυτές δεν έλαβαν τη δέουσα προστασία από το κράτος. Να αναφέρω μία από τις αναδυόμενες τάσεις που βλέπουμε όλο και περισσότερο. Μία αύξηση όσον αφορά τις εκστρατείες δυσφήμισης προκειμένου να σπηλωθεί ουσιαστικά η υπόλοιψή τους, να θεωρηθεί παράνομη και παράτυπη η δραστηριότητά τους, δέχονται συνεχώς απειλές στα πλαίσια μιας εκστρατείας δυσφήμισης που τους παρουσιάζει ως προδότες, ως πολέμιους του κράτους, ως κατασκόπους, ως ξένους πράκτορες ή γενικά ως πολέμιους της ανάπτυξης. Επομένως, κατά αυτόν τον τρόπο δεν δέχονται μόνο ατομικές επιθέσεις, αλλά νομιμοποιείται κατά κάποιον τρόπο μία επίσημη θεσμική επίθεση που γίνεται εναντίον τους. Υπάρχει μια κινητοποίηση, αν θέλετε, της κοινωνίας ή ακόμα και του κράτους των θεσμών εναντίον τους. Οι εκστρατείς αυτές της φήμησης και σπήλωσης γίνονται πολλές φορές και μέσω των μέσω μαζικής ενημέρωσης, γίνονται επιγραμμικά στο διαδίκτυο και μπορούν να οδηγήσουν σε πολλές σωματικές επιθέσεις. Στην Τανζανία, για παράδειγμα, πέρυσι, μετά από μια ευρεία τέτοια εκστρατεία σπήλωσης κατά της κοινότητας ΛΟΑΔ, παράδειγμα, οι υπερασπιστέ τη κοινότητα αυτή δέχθηκαν πολλέ απειλέ, αλλά ακόμα και σωματικέ επιθέσει. Να φορέσει και τα ακουστικά της η Γιολάντα για να ακούει τα όσα λέμε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις οι οποίες παραβιάζουν οι ίδιες τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το βλέπουμε αυτό σε αυθαίρετες συλλήψεις, στην άσκηση βία, στα βασανιστήρια, που αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό της, της τάξη του 63% όσον αφορά όλα αυτά τα φαινόμενα βίας. Βλέπουμε ότι πολύ συχνά ένα 27% των κατηγοριών έχουν να κάνουν με την κατηγορία της διατάραξης δημόσιας τάξης ή την κατηγορία των παράνομων δημόσιων συγκεντρώσεων, αλλά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο κατηγορούνται για παραβάσεις ε, οι οποίες μπορούν αυτή τη στιγμή να τιμωρηθούν και με κάθριξη, όπως για παράδειγμα 32 χρόνια κάθριξη για έναν ακτιβιστή στο Μπουρούντι ο οποίος κατηγορήθηκε για εξέγερση ή για την καταπάτηση του κράτους δικαίου ή επειδή είχε στραφεί κατά της θαντικής ποινής. Υπάρχουν και συγκεκριμένε νομοθεσίε οι οποίε αποτελούν αντικείμενο κατάχρηση προκειμένου να στραφούν κράτη εναντίον των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπω για παράδειγμα μια νέα αντιτρομοκρατική νομοθεσία στην Ικαράγουα, στα πλαίσια τη οποία πλέον μπορεί να κατηγορηθεί για τρομοκρατία ακόμα και κάποιο ο οποίο κατηγορείται για την ζημία κατά ακίνητη περιουσία. Καταλαβαίνετε, οποιοδήποτε ουσιαστικά μπορεί να κατηγορηθεί για κάτι τέτοιο. Στον Μπαγκλαντέ έχουμε ένα νέο νόμο όσον αφορά την ψηφιακή ασφάλεια. Εδώ πέρα θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα και ποινέ 14 τεσσάρων ετών για οποιονδήποτε προκαλεί οποιαδήποτε ζημία στο κράτος μέσω του διαδικτύου. Καταλαβαίνετε ότι πάλι η κατηγορία είναι ιδιαίτερα γενική και μπορεί οποιοδήποτε να βρεθεί να κατηγορείται για το παράπτωμα αυτό. Επίσης, στα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουμε κάποιες νέες νομοθεσίες όπου βλέπουμε ότι ο Αχμέτ Μανσούρ καταδικάστηκε σε δεκαετή κάθερξη για κατηγορίες σε σχέση με την διάδοση ψευδών ειδήσεων επιγραμμικά και κατά αυτόν τον τρόπο για το ότι στράφηκε κατά της υπόλοιψης του ίδιου του κράτους. Τώρα, για ποιο λόγο θα πρέπει να περασπιζόμαστε τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επειδή έχουμε ουσιαστικά πάρα πολλά θετικά επιτεύγματα και επειδή έχουμε σημειώσει ήδη μια πάρα πολύ σημαντική πρόοδο στην προάσπισή τους βλέπουμε ότι όλες αυτές οι προσπάθειες καταστολής που λαμβάνουν χώρα είναι μια αντίδραση τελικά στο ότι αυξάνεται η δράση και αποτελεσματικότητα των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη Μαλαισία, για παράδειγμα, οδηγηθήκαμε σε ένα μορατόριμο όσον αφορά την θανατική ποινή, άλλαξε ουσιαστικά η στάση τη κυβέρνηση. Στη Λατινική Αμερική, οι υπερασπιστέ αυτοί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οδήγησαν στην συμφωνία μια, στην σύναψη μια συμφωνία στην οποία συμμετέχουν 24, διαφορετικές, 24 διαφορετικά κράτη της Λατινικής Αμερικής, ενώ στο Κονγκό μετά από πάρα πολλά χρόνια και μετά από την έντονη δράση γυναικών υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλο και περισσότερε γυναίκε μπορούν να έχουν πλέον τη δική του γεωργική εκμετάλλευση. Σα έχω μοιράσει κάποια φυλάδια τα οποία περιγράφουν τι μπορείτε να κάνετε εσεί ω βουλευτέ για να προασπίσετε του υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περιγράφουμε το έργο του και κάνουν και κάποιες συστάσεις σε εσά για το πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε τους ανθρώπους αυτούς από το αξίωμα το οποίο έχετε. Αυτά όσον αφορά την παρουσίασή μου και είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω τυχόν ερωτήσει. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πραγματικά την τύχη να έχουμε μαζί μα δύο αυτόπτε μάρτυρες, δύο υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έρχονται από δύο διαφορετικέ περιοχέ. Η Γιολάντα Περέ Κρούστα θα πάρει πρώτα τον λόγο, η οποία συμβολίζει και εκπροσωπεί όλο αυτό τον αγώνα που δίνουν οι αυτόχθονοι πληθυσμοί για να προασπίσουν το δικαίωμά τους ε, στην ε, ιδιοκτησία και η οποία θα αναφερθεί επίσης και στην αυθαίρετη σύλληψη ε, του συζύγου της, ο οποίος ήταν και αυτός αυτόχθον υπερασπιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ας δώσουμε λοιπόν καταρχάς το λόγο στην πρώτη καλεσμένη μας, τη Γιολάντα. Καλημέρα σας, ε, βουλευτές. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Frontline για την ε, πρόσκληση, καθώς επίσης και όλες τις οργανώσεις, παν συντονιστικό από τη Γερμανία, την ε, πολιτική υπηρεσία για την ειρήνη και άλλες υπηρεσίες και άλλες ΜΚΟ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε για το χώρο που μου ανοίγετε για να μπορέσω να μιλήσω, να μ' ακούσετε να ακούσετε τα δεινά που υποφέρουμε στο Μεξικό. Λέγομαι Γιολάντα Πέρες Κρούς. Είμαι σύζυγος του αγωνιστή Πάμπλο Λόπες Αλαβές. Είμαι και εγώ αγωνίστρια και υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατάγομαι από το Σάνι Σίδρο Αλοάπαμ. Η γλώσσα μου λέγεται Σαποτέκο από το βουνό Σχέρα Χοάρες και την πολιτεία Ουαχάκα του Μεξικού. Για ποιο λόγο αγωνίζομαι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς αυτόχθονες λέει, υπερασπιζόμαστε τη φύση της μάνας γης, το νερό μας, τα ζώα του δάσους. Αυτό υπερασπιζόμαστε και προασπίζουμε. Αλλά επειδή έχουμε μια κυβέρνηση ε, που είναι πραγματικά ε, υποστηρίζουν ε, αυτούς που θέλουν να εκμεταλλεύονται το δάσος. Δεν τους ενδιαφέρει ε, ούτε το νερό, ούτε η φύση, ούτε η μάνα γη. Γι' αυτό το λόγο μας φυλακίζουν. Μας φυλακίζουν άδικα. Μας απαγάγουν και μας κρατούν ομήρους, μας θανατώνουν, επειδή υψώνουμε τη φωνή μας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήρθα να σας μιλήσω για την περίπτωση του συζύγου μου, Πάμπλο Λόπες Σαλαβές, ο οποίος είναι ηθαγενής της φυλής των Σαποτέκ. Από το 2010 τον έχουν απαγάγει και τον κρατούν φυλακισμένο. Μέχρι σήμερα άδικα. Για το λόγο αυτό αναγκάστηκα να αφήσω το σπίτι μου. Αναγκάστηκα να αφήσω ό,τι έχω και δεν έχω, τα υπάρχοντά μου στο χωριό μου. Και να φύγω από τη χώρα για να απαιτήσω δικαιοσύνη, για να απαιτήσω να αφαιθεί ελεύθερος ο σύζυγός μου. Διότι εγώ ξέρω τι άνθρωπος είναι ο σύζυγός μου. Εγώ ξέρω ότι τον κατηγορούν για εγκληματία. Ποινικοποιούν τη δράση του. Πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση να παραβιάζει έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματα των αυτοχθόνων ηθαγενών λαών. Πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση του κράτους της Μεξικανικής Δημοκρατίας να υποβάλουν σε τέτοια δεινά τους αυτόχθονες ηθαγενείς. Γι' αυτό το λόγο έφυγα από τη χώρα και βγήκα να ψάξω κόσμο, ταπεινούς ανθρώπους όπως είστε εσείς, για να με υποστηρίξουν. Για να με στηρίξουν. Για να απαιτήσω να τηρηθεί η απόφαση 23 κάθετος 2017, 23 κάθετος 2017 της ομάδας εργασίας για την αυθαίρετη κράτηση. Είναι μια ομάδα εργασίας του ΟΗΕ αυτή. Ε, υπό ποια έννοια. Να αφαιθεί αμέσως ελεύθερος ο σύζυγός μου Πάμπλο Λόπες Λαβές και να αποζημιωθούν να αποκατασταθούν οι ζημίες. Εννιά χρόνια τον έχουν στη φυλακή. Άδικα. Πώς είναι δυνατόν να με απειλούν ότι θα με σκοτώσουν επειδή απαιτώ να αφαιθεί ελεύθερος ο σύζυγός μου. Πώς είναι δυνατόν τα παιδιά μου να μην βλέπουν τον πατέρα τους. Πώς είναι δυνατόν να παραβιάζονται έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Της οικογένεια μου, τα δικά μου, των παιδιών μου. Πώς είναι δυνατόν. Να είμαστε χωρισμένοι με την οικογένειά μου. Σας παρακαλώ να απαιτήσετε και εσείς την άμεση απελευθέρωση του συζύγου μου. Πάμπλο Λόπες Αλαβές. Και σας ευχαριστώ πολύ. για την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλους σας και κάθε ένα ξεχωριστά που ακούτε τον πόνο μου τα δεινά που μας επιβάλλει η κυβέρνηση. που μας επιβάλλει η κυβέρνηση, λέω, του Αλεξάνδρου Μωράτ. Και ελπίζω ότι η μεξικανική κυβέρνηση θα με υποστηρίξει τελικά και θα αφήσει ελεύθερο το σύζυγό μου. Πάμπλο Λόπε Αλαβέ. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ, Ιολάντα. Αυτή η μαρτυρία είναι πάρα πολύ συγκινητική, ε, αλλά πάρα πολύ ε, ενδεικτική και εύγλωτη για τον αγώνα των αυτοχθόνων λαών που αγωνίζονται για το κλίμα, τη βιοπικιλότητα, θέματα ιδιοκτησίας της γης. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη μαρτυρία. Τώρα θα δώσω το λόγο σε έναν εκπρόσωπο από την Κυργυζία, τον Αμπτούλ Χαλίλοφ, ο οποίος είναι ο συνήγορος του κυρίου Ασκάροφ, εξέχοντα ε, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κυργυζία. 20 χρόνια εργαζόταν εκεί προς την κατεύθυνση αυτή πριν το συλλάβουν και τον φυλακίσουν το 2010. Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε ότι έχει καταδικαστεί σε ισόβια στην Κυργυζία. Θα σας δώσω αμέσω το λόγο για να μας εξηγήσετε πώς έχει σήμερα η κατάσταση. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το όνομά μου είναι Σερτομπέκ. Είμαι δικηγόρος για την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εδώ ήθελα να παρουσιάσω την υπόθεση του Αζιμτζάν Ασκάροφ ενός γνωστού ε, ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το Κυργιστάν. Ε, τον Ιούνιο του 2010 υπήρχαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των Κυργίζιων και των Ουσμπέκων στο νότιο Κυργιστάν. 400 ε, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τρεις μόλις μέρες. Πριν από τη σύλληψή του, ο κύριος Ασκάροφ είχε δει ότι υπήρξε λαϊλασία, εμπρισμός και βίες επιθέσεις ε, λόγω αριθμητικών διαφορών στην ε, γενέτειρά του, στην πόλη από την οποία προέρχεται. Η, ε, είχε μάλιστα κινηματογραφήσει, είχε βιντεοσκοπήσει τέτοιες σκηνέ πριν τον συλλάβει αστυνομία. Ε, συνελήφθη τον Ιούνιο του 2010 επειδή υποτίθεται ότι εκείνος ήταν υποκινητής μαζικών ε, διαδηλώσεων και υποκίνησε και ε, διαφορετικό ε, μίσους στην ε, περιοχή του. Οι συγγενείς μάλιστα του ίδιου του κυρίου Ασκάροφ δέχτηκαν απειλές και, σωματική, και απειλές σωματικής βίας και κατά τη δίκη του ο κύριος Ασκάροφ ε, ε υπερασπίστηκε με βάσιμα επιχειρήματα την υπόθεσή του αλλά ο εισαγγελέα αρνήθηκε τι επανειλημμένε εφέσεις του ε, από τη στιγμή που μπήκε στη φυλακή. Η ακρόαση, μάλιστα η δημόσια ακρόαση, έγινε σε ατμόσφαιρα μίσους όπου συγγενείς του νεκρού αστυνομικού ε, φώναζαν βρισχές κατά των ε, Ουσμπέκων καθώς και προσβολές και ζητούσαν την άμεση τιμωρία από την πλευρά των δικαστικών λειτουργών ή των αστυνομικών. Ήταν σαφέ στη διάρκεια τη ακρόαση ότι ο κύριο Ασκάροφ είχε δεχτεί ξύλο δαρμό και κατά πάσα πιθανότητα στην κράτησή του είχε υποβληθεί και σε βασανιστήρια. Τον Σεπτέμβριο του 2010 ο Ασκάροφ και κάποιοι άλλοι βρέθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν σε ισόβια. Το 2012, αφού εξάντλησε όλα τα ενδικά μέσα σε εθνικό επίπεδο, οι δικηγόροι του υπέβαλαν έτοιμα ενώπιον της ε, Επιτροπής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Μάρτιο του 2016 η Επιτροπή αυτή κατέληξε ήταν παράνομη η κράτηση του κυρίου Ασκάροφ σε απάνθρωπες συνθήκες με βασανιστήρια και κακομεταχείριση ε, χωρίς το δικαίωμα σε μία νόμιμη δίκη. Η Επιτροπή κατέληξε ότι το Κυριζιστάν πρέπει να αναλάβει τα απαραίτητα βήματα, δράση για να απελευθερωθεί ο Ασκάροφ και να καταργηθεί η καταδίκη του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τις αρχές του Κυργιζιστάν να εφαρμόσουν τις συστάσει της Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βάσει της απόφασης της Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το δικαστήριο αποφάσισε να ξαναδεί την υπόθεσή του. Άρχισαν να υπάρχουν κάποιες ε, ελπίδες, αλλά τον, ε, ε, το 2018 το Μάρτιο τελικά επαναλήφθηκε η ποινή του και η καταδίκη του και παραμένει στη φυλακή. Ο κύριος Ασκάροφ μέσω όλων των, ε, ε, ανθρωπίνων, των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητά να απελευθερωθεί μαζί με όλους τους συγκρατουμένους του. Στις 18 Μαρτίου 2019, στα πλαίσια της συνολικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωκοινοβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επανεξέταση της ε, ποινή ε, του κυρίου Ασκάροφ και ζήτησε να απελευθερωθεί αμέσως καθώς και να του πληρωθεί αποζημίωση. Όπως είπα, η υπόθεση του κυρίου Ασκάροφ είναι η φέστατη απόδειξη της ε, πλήρους αδικίας που επικρατεί στο νότιο Κυργιζιστάν λόγω των εθνοτικών συγκρούσεων κατηγορία, η άδικη κατηγορία και η άδικη εκδίκαση των υποθέσεων των Ουσβέκων δείχνουν ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση από τις ένομες δυνάμεις, ε, αστυνομικούς και δικαστές κατά των Ουσβέκων, χωρίς έρευνα με απευθείας διώξεις και με δυσανάλογη στόχευση της ουσμπεκικής μειονότητας. Αυτό έχει οδηγήσει σε καταδίκες και εισόδια πολλές φορές. Ο κύριος Ασκαρόφ είναι ένας από τους 54 ουσμπέκους που βρίσκονται στη φυλακή. Το Μάρτιο του 2019 ο κύριος Ασκαρόφ μεταφέρθηκε σε μια ειδική φυλακή την λεγόμενη, το λεγόμενο στο τόπο εδώ υπαριθμό 19, με ειδικό καθεστώς. Ο κύριος, η υγεία του κύριου Ασκαρόφ έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ και όλα του τα περιουσιακά στοιχεία έχουν παγώσει ε, μεταξύ των οποίων και το σπίτι του. Σήμερα θέλω λοιπόν να εκφράσω την ε, έντονη ανησυχία μας για την άδικη και συνεχιζόμενη φυλάκιση του Αζίμοφ ε, Ασκάροφ, Αζίμον Ασκάροφ, καθώς και την επιδείνωση της υγείας του. Σας καλώ να απευθύνετε έκκληση στην κυβέρνηση της Κυργυζίας για να τον απελευθερώσει αμέσως και να κάνει ό,τι μπορεί για εκείνον. Ε, θα πρέπει να απελευθερωθεί ο κύριος Ασκάροφ, να λάβει ιατρική ε, βοήθεια και να μπορέσει να ξαναβρεθεί με την οικογένειά του σε ένα ασφαλέ περιβάλλον. Εκ μέρου του κυρίου Σκάροφ και τη οικογένειά του, σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Εάν έχετε ε, κάποια ερώτηση, είμαστε στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα περάσω απευθεία στην Λάουρα Μπατιστίν υπεύθυνη της γραμματείας του Protect Defenders. Ε, έχετε το λόγο. Thank you very much for this. Σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα αυτή που μου δίνετε να κάνω την παρουσίαση αυτή. Είδαμε κάποια εμβληματικά παραδείγματα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση περασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διεθνής κοινωνία των πολιτών, καθώς επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει αδιαφορήσει απέναντι στις προκλήσεις και τις δυσκολίες αυτές. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω σήμερα τον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που φέρει το όνομα protectdefenders.eu. Το θεσπίστηκε ο μηχανισμός αυτός και έχει ως στόχο να προασπίσει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν τους υψηλότερους κινδύνους και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εφαρμάζεται από μια κοινοπραξία 12 οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μέσω του προγράμματος αυτού καταφέρνουμε να έχουμε μια πλήρη υποστήριξη όχι μόνο σε μεμονωμένους ακτιβιστές, αλλά και σε τοπικές οργανώσεις και σε τοπικές κοινότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ProtectDefenders.eu έχει ως στόχο να βοηθήσει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περιοχές του κόσμου που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να υπερασπίζεται κανείς τα ανθρώπινα δικαιώματα και επικεντρωνόμαστε σε ακτιβιστές, σε υπερασπιστές που αποτελούν στόχο απειλών, όπως για παράδειγμα οι περιπτώσεις που ακούσαμε πριν από λίγο, άνθρωποι οι οποίοι υπερασπίζονται τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΔΜΑ, τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Αναφερόμαστε επίσης σε δικηγόρους, σε όσους υπεραμείνονται της ελευθερίας της έκφρασης ή της θρησκευτική ελευθερίας. Θα ήθελα πολύ σύντομα να σας δώσω κάποια παραδείγματα σε σχέση με τα επιτεύγματα τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Μέσω του προγράμματος λοιπόν αυτού καταφέραμε να χορηγήσουμε περίπου 1.293 επίγουσες επιδοτήσεις σε 1.700 περασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τους υποστηρίξαμε δηλαδή προκειμένου να έχουμε μία επίγουσα με την κατάστασή τους, προκειμένου να τους προσφέρουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δικηγορική υποστήριξη, να τους επανενώσουμε τις οικογένειές τους κ.ο.κ. Υποστηρίζουμε 100 85 τοπικές ε, οργανώσεις στις προσπάθειές τους να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, μολονότι λειτουργούν σε ένα πολύ αντίξω περιβάλλον και μολονότι ο ζωτικό του χώρο ε, συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο. Πάνω από 600 υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουμε βοηθήσει να μετεγκατασταθούν σε ασφαλείς τόπους ενώ αντιμετωπίζουν άμεσες απειλέ ή ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο. Οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν να, να μετεκατασταθούν ε, ενδεχομένως στο στερικό της χώρας τους, σε μια κάποια άλλη περιφέρεια, σε μια άλλη περιοχή ή ακόμα και σε κάποια άλλη χώρα. Οι περισσότερες από τις ε, μετεκαταστάσεις αυτές που έχουμε εμεί παράσχει διευκολύνονται μέσω μιας πλατφόρμας. Μια πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν πάνω από 60 μέλη, όπου συμμετέχουν ε, δήμοι, πανεπιστήμια, περιφερειακές κυβερνήσεις, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, που ουσιαστικά έχουν προγράμματα υποδοχής ε, και συγκεκριμένα καταφύγια για αυτούς τους ε, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλές φορές δραστηριοποιείται η ίδια η κυβέρνηση, Υπουργοί Εξωτερικών, τοπικές κυβερνήσεις, όλοι αυτοί συμμετέχουν σε αυτή την πλατφόρμα που έχουμε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε μια θετική και γόνιμη ανταλλαγή θετικών πρωτοβουλειών που έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόσουν ορισμένα κράτη υπέρ των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα έλεγα ότι μία από τις πιο σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι το πώς θα καταφέρουμε να διευκολύνουμε τη χορήγηση θεωρήσεων για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άνθρωποι οποίοι αντιμετωπίζουν έντονους κινδύνους και επιγόντως πρέπει να μεταβούν σε κάποια άλλη χώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για μας να έχουμε αυτόν τον θετικό διάβλο επικοινωνίας με τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία ενεργά υποστηρίζουν το πρόγραμμα αυτό για την υπεράσπιση, των για την υπεράσπιση και την προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίση, παράσχουμε προγράμματα κατάρτιση και εκπαίδευση, καθώ επίση και προγράμματα ευαισθητοποίηση, εκστρατείε ενημέρωση και μπορείτε να δείτε περισσότερε λεπτομέρειε στο φυλάδιο αυτό το οποίο σα διανύμαμε. Ωστόσο θα ήθελα να αφιερώσω τα τελευταία αυτά δύο λεπτά της παρουσίασής μου σε κάποια νέα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει. Όπως σας είπα, ο μηχανισμός αυτός ανανεώθηκε, επικαιροποιήθηκε για τα επόμενα τρία χρόνια και προκύπτουν αυτή τη στιγμή κάποιες νέες προκλήσεις, οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ακούσαμε ότι πολλοί υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν έντονε δυσχέρειε και αντικσότητε, αλλά από την άλλη θα έλεγα ότι ουδέποτε το κίνημα υπερίσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν ήταν τόσο ευρύ και τόσο παγκόσμιο όσο είναι τώρα. Και από τότε που έγινε η διακήρυξη για την υπεράσπιση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν από 20-21 χρόνια, έχουμε δει ότι έχει αυξηθεί σημαντικότατα ο αριθμό των ίδιων των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δράσεις τους αυξάνονται παντού, αλλά εξακολουθούν και αποτελούν βέβαια θύματα απειλών, δολοφονιών, αυθαίρετων συλλήψεων και κρατήσεων. Και ας μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι επιθέσεις βασίζονται σε, μια, σε ένα διάχυτο αφήγημα που τους παρουσιάζει ως εχθρούς των κρατών, ως τρομοκράτες. Αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο όπως είπατε, είναι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι υπερασπίζονται τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, τα δικαιώματα στη χρήση της γης, οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών, αυτοί που υπερασπίζονται τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΔΜΑ και αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο απομονωμένοι, αυτοί που βρίσκονται στις πιο απομακρυσμένε περιοχές. Λαμβάνοντα λοιπόν υπόψη το νέο αυτό πλαίσιο και τις νέες αυτές προκλήσεις, τα επόμενα τρία χρόνια θα επικεντρωθούμε πάρα πολύ στο να καταφέρουμε να έχουμε μια προσέγγιση υπεράσπισης που να λαμβάνει υπόψη την ισότητα των φύλων. Θέλουμε να καταφέρουμε να αποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες των υπερασπιστών αυτών που προασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με αυτού που βρίσκονται σε απομονωμένε περιοχέ, που βρίσκονται μακριά από τι πρωτεύουσε των χωρών του, εκεί που δεν υπάρχει πραγματικά δίκτυο τη διεθνή κοινότητα που θα μπορούσε να του εντοπίσει και να του προστατεύσει. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται για να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την δική σας την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όλους τους ευρωβουλευτές, ευρωβουλευτές που έχουν υποστηρίξει τα τελευταία χρόνια τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο από πολιτικής πλευράς για κάποια ευαίσθητα ζητήματα, αλλά και όλους όσους έχουν προσπαθήσει να προωθήσουν περισσότερο το έργο μας και να χρηματοδοτήσουν περισσότερο τα προγράμματα προστασίας των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προφανώς θέλουμε να συνεχίσουμε την γόνιμη αυτή συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες ή για να εμβαθύνουμε σε επιμέρους ζητήματα τα οποία ενδεχομένω να σας ενδιαφέρουν. ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στους βουλευτές. Η κυρία Σάντους βλέπω να ζητά το λόγο ήδη. Χαιρετώ την κυρία Γιολάντα Πέρες Κρούς η οποία μας ε, έχει δώσει μια πολύ γλαφυρή μαρτυρία του τι συμβαίνει στη χώρα της και με τους ε, ηθαγενείς εκεί. Θα μιλήσω τώρα πορτογαλικά. Ήθελα να χαιρετήσω τους δύο ακτιβιστές. Γνωρίζω πολύ καλά τις περιπτώσεις τους, διότι επί οκτώ χρόνια παρακολουθούσα πολύ καλά το τι συμβαίνει στις περιοχές σας και γνωρίζω και τα γεγονότα. Οι Ουσμπέκοι κινδυνεύουν στο Κυρκίζιστάν ή Κυργιζία. Η Κυργιζία. Η δίωξη των Ουσμπέκων, που είναι μειονότητα, πρέπει να μας ανησυχεί. Η περίπτωση που αναφέρεται εδώ, η δίκη αυτή αφορά όλους τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρά τις επιταγές των διεθνών δικαστηρίων, ε, το κράτος, το κρατικό δικαστήριο, το κρατικό δικαστικό σύστημα εμένει. Εμένει στην κράτηση αυτών των ανθρώπων. Όμως τα λόγια μου και οι ερωτήσεις μου θα έπρεπε να σας καθησυχάσουν, γιατί θεωρούμε ότι δεν ήρθατε εδώ εις Δεν θα πέσουν στο κενό αυτά που μας είπατε. Όλοι εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε για τη διάσωση των ανθρώπων αυτών. Και εδώ δεν θέλω να θέσω ερωτήσεις στους δύο προσκεκλημένους μας. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να προασπιστούμε το ρόλο σας. Και ο ρόλος σας ε, μπορεί να διαφυλαχθεί καλύτερα χωρίς να θέτουμε άλλα ερωτήματα, αλλά απλώς να ακούμε τα γεγονότα όπως τα παρουσιάσατε και τα εκθέσατε. Τώρα για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και για το μηχανισμό που εσείς χρησιμοποιείτε. Είναι πολύ καλή η δουλειά σας, είναι πολύ θετικό το αποτέλεσμα πιστεύω και πολύ διεξοδικό ο τρόπος που εργάζεστε, πολύ επιστημονικός, αλλά για τις απειλές κατά των ακτιβιστών. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει πολλά ακτιβιστές και χειροτερεύουν τα πράγματα. Τον μηχανισμό λοιπόν αυτό, πώς θα τον επικυρωποιήσετε τα ερχόμενα χρόνια για να μπορούμε να δώσουμε μια απόκριση προσαρμοσμένη στις στις σημερινές ανάγκες καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες που παρουσιάζονται στην πράξη, κάνοντας μια αξιολόγηση από την εφαρμογή του μηχανισμού σήμερα. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο μηχανισμός τα ερχόμενα χρόνια και ποιοι είναι οι δικοί σας στόχοι στην ε, χρήση του μηχανισμού αυτού και τι υποστήριξη θα θέλατε να λάβετε. Ευχαριστούμε. Πόλντο. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον πόνο της Γιολάντας και του Παύλο. Έχω ένα γιο, ο οποίος καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση. Πέντε χρόνια έχω να τον δω. Πέντε χρόνια είμαι εξόριστο στη χώρα μου. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι μακριά από την οικογένειά σου και ξέρω τι σημαίνει να είσαι μακριά από τον νόμο και ξέρω ότι ε, ε, σημαίνει να είσαι ανυπεράσπιστος απέναντι στον νόμο. Μπορείτε να, υποστηρί... να προσβλέπετε στην υποστήριξή μου και όλων των βουλευτών. Έχω να ρωτήσω κάτι. Όταν μιλάμε για τις χώρες που κινδυνόβουν περισσότερο, προηγουμένως μιλήσαμε για Κολομβία, Μεξικό, Βραζιλία και Φιλιππίνες στο προηγούμενο θέμα. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν αναφερθήκαμε σε χώρες όπως είναι η Κούβα, η Βενεζουέλα, η Νικαράγουα. Πώς ορίζονται οι υπερασπιστές, οι αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσύ πώς τους ορίζετε, πώς υποστηρίζουμε εκείνους που πέφτουν νεκροί στις διαδηλώσεις από τη βίαιη καταστολή των κυβερνήσεων. Για ποιο λόγο δεν μπαίνουν σε αυτή την ιεράρχηση, τη λίστα των χωρών, για να μην μιλήσω για άλλες χώρες, όπως είναι φυσικά η Κορέα, η Κίνα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, εσάς τους υπερασπιστές και αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους υπερασπιστές των υπερασπιστών, ποια είναι τα κριτήρια σας για να κάνετε αυτή την ιεράρχηση. Γιατί αισθάνομαι λίγο εγκαταλελειμμένος. Γιατί δεν υπερασπιζόμαστε αυτούς που υπερασπίζονται το κράτος δικαίου ως πρώτη αξία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κάθριν Χάουιτ. Uh, uh, Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση στους frontline γιατί είπατε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ε, δολοφονιών ε, των ακτιβιστών έχει να κάνει με περιβαλλοντικά δικαιώματα, δικαιώματα ηθαγενών και δικαιώματα για τη, στην γη, στο χώρο που διαμένουν. Ε, ελπίζουμε ότι τα ότι οι θύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν ενσωματώσει αυτά στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δουν τι μπορούν να βελτιώσουν. Τώρα για, την προστασία, για τους protect defenders. Ήθελα να μας πείτε τι προκλήσεις αντιμετωπίζετε τι δυσκολίες όταν θέλετε να πάρετε θεωρήσεις ε, σύντομης διάρκειας και αν εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την χορήγηση ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Μπορεί κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ πέρα. Ευχαριστούμε. Ιρέν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλος ιδιαιτέρως την κυρία Πέρες Κρούς που ήρθες εδώ. Με συγχωρείτε, δεν βλέπω το όνομά σας από εδώ. Και τον κύριο Αντράλιλοφ που ήρθες εδώ. Για τον κύριο Αντχάλιλοφ έχω λοιπόν ερωτήσεις. Και εγώ είμαι δικηγόρος, ε, ως δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, πώς βλέπετε ακριβώς το ρόλο των δικηγόρων θεωρείτε ότι χρειάζεται περισσότερο, ότι και εσεί ο ίδιο θα θέλατε να λάβετε προστασία ω συνήγορο κάποιου ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσεί δεχτήκατε προσωπικώ απειλέ, επειδή είχατε αυτού του πελάτε. Και τι μπορούμε εμεί να κάνουμε συγκεκριμένα για να ενθαρρύνουμε περισσότερου δικηγόρου να γίνουν περασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είτε με κάποιο ειδικό, κάποια ειδική αμοιβή, πώ μπορούμε να του προστατεύσουμε. Ευχαριστούμε. Άννα. Καταρχάς, ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πέρεσκους και τον κύριο Αυτολαχή ε, για την, ε, την παρουσία τους εδώ και τις ιστορίες που μας παρουσίασαν. Για μένα είναι πάντοτε πολύ εμψυχωτικό να ακούω το θάρρος και την τόλμη που δείξατε. Στη δική μου χώρα τα δικά μας εκλογικά αποτελέσματα ήταν πολύ καλά ακριβώ χάρη στη δράση ακτιβιστών. Πώς εγώ θα μπορούσα να κοιμάμαι ήσυχη, ξέροντας ότι άνθρωποι σαν και εσάς που έχουν προσφέρει τόσα πολλά δέχονται απειλές για τη ζωή, κατά τη ζωή τους. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, και εγώ από τη δική μου πλευρά για τη χώρα, εκ της χώρας μου, όπου έχουμε αντίστοιχα προβλήματα και έχετε εμπνεύσει ανθρώπους σαν και εμένα. Ε, και τώρα να κάνω και μια ερώτηση και για τους frontline defenders ίσως. Ξέρω ότι έχετε ένα πολύ καλό δίκτυο, αλλά κάποια στιγμή φαίνεται να μην υπάρχει άλλη λύση παρά την ε, ε απομάκρυνση των ανθρώπων αυτών και τον εκτοπισμό τους. Να ζήσουν αλλού δηλαδή. Πού θα πρέπει να πηγαίνουν οι ακτιβιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να έρθουν κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάπου αλλού κοντά στην περιοχή του, στην περίπτωση τη επαναγκατάσταση. Γιατί Εάν ε, δεν κάνουμε κάτι εδώ, τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε κύριο Σκουλόκλου. Um, θα ήθελα να συγχαρώ και τους δύο προσκεκλημένους μας, τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και ε, εκείνους που υποφέρουν από την καταστολή στις χώρες αυτές. πολύ εύστοχα επιλέξατε χώρες όπως είναι η Κολομβία, όπου κάθε μέρα δολοφονείται και κάποιος και στις άλλες χώρες, στο Μεξικό και τις Φιλιππίνες. Η τέταρτη ποια ήταν, δεν θυμάμαι. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην καταστολή και τις δελοφονίες και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαφθορά των κυβερνήσεων στις χώρες αυτές που αναφέρατε. Υπάρχει σχέση. Ευχαριστώ. Ήθελα απλώ να πω ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις μαρτυρίες σας, ευχαριστώ για τη δουλειά σας και τον αγώνα σας. Ήθελα απλώς να πω ότι οπουδήποτε και αν σκεφτεί κανείς τη γη, τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και μπορεί να δέχονται πιέσεις ή επιθέσεις, όπου και αν συμβαίνει αυτό πρέπει να το λέμε και να το φωνάζουμε. Είμαι υπεύθυνη εισηγήτρια για την έκθεσή μας εδώ, για την κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίω, για την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε, σε σχολιασμό της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2018 και ω συνέχεια της δικής μας Επιτροπής από το 2018 επίσης, για όλα αυτά που γίνονται, που κάνετε εσείς, που κάνουμε εμείς, Όλα είναι απαραίτητα. Δεν υπάρχει τίποτα το περιττό. Και πραγματικό ευχαριστώ, πραγματικά ευχαριστώ για όλους τους ακτιβιστές παντού στον κόσμο. Αναφέρθηκε εδώ και ο μηχανισμός Defenders EU. Εάν υπάρχει κάτι παραπάνω που μπορούμε να προσφέρουμε για το μηχανισμό αυτό, μην διστάσετε να μας το ζητήσετε. Θα επιληφθούμε. Ο κύριος Μπάνιον. Ναι, είχα ακόμα τα ακουστικά μου για να ακούσω την κρυμμηνία. Σε ποιο βαθμό οι προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επαναπατρίζονται, επανεγκαθίστανται, σε τι βαθμό μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Διότι στην εποχή μας πολλά μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά, στο ίντερνετ. Δεν χρειάζεται να είναι κανεί μέσα στη χώρα όπου θέλει να περασπιστεί τα δικαιώματα. Μπορεί να είναι μια λύση λοιπόν να του απομακρύνει κανεί από τη χώρα όπου αρχικά έκαναν τη δουλειά και παρόλα αυτά να μπορούν ενεργά να προσπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή. Υπάρχει τέτοια του είδου τάση. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να θέσω μια ερώτηση στην, ε, ε, στην εκπρόσωπο του Human Rights Defenders. Είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε ανθρώπους που τους ε, φέραμε στην Ευρώπη με θεωρήσεις. Ανθρώπους που δέχονταν απειλές και στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια από τη διασπορά των χωρών τους, από τους ε, μετανάστες των χωρών τους και από μηνύματα της χώρας προέλευσης ε, ακτιβιστέ Τούρκοι λόγω χάρη που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Ευρώπη, οι οποίοι δέχονται απειλέ με μηνύματα απευθεία από την κυβέρνηση τη Τουρκία. Έχουμε επίση τη λεγόμενη ρωσική διασπορά, του Ρώσου μετανάστε, που μπορεί να απειλεί ή να εκτοξεύει απειλέ κατά των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη τώρα. Ε, τι γίνεται με του ακτιβιστέ αυτού λοιπόν που βρίσκονται στην Ευρώπη και συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν και στη χώρα του ή τέλο πάντων συνεχίζουν να φέρνουν ει πέρα στα καθήκοντά του για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δίνω το λόγο σε εκείνους που αφορούσαν ε, οι ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις. Χαίρομαι που δείξατε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε συστηματικά διάλογο. Ως προς την προσωρινή επαναγκατάσταση, η μεταγκατάσταση, μπορεί να χρειαστεί μόνο για κάποιους μήνες. Τη στιγμή που βρίσκεται σε όξενση ...ή ε, σύγκρουση ή που οι πιέσει είναι πολύ ψηλέ. Μετά μπορεί να γυρίσει κανεί στη χώρα και να συνεχίσει τη δουλειά του. Το σύστημα που σας εξήγησα ξεκινάμε μια τρίμηνη κλασική θεώρηση και νομίζω ότι το πιο, ε, το πιο το πρόγραμμα που καλύπτει καλύτερα είναι διετές ε, για συγγραφείς, ε, ανθρώπους που δραστηριοποιούνται και γραπτός. Η Γάλλοι άρχισαν να στηρίζουν το πρόγραμμα αυτό και όταν είδαν ότι η ΕΔΟ δεν μπορεί να βοηθήσει, ε, μπορούν να στηρίξουν το πρόγραμμα αυτό. Οι ακτιβιστές όμως συνήθως είναι πολύ ε, παθιασμένοι, δεν θέλουν με, το σκοπό, με τον αγώνα τους, δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα, δεν θέλουν να φύγουν. Πολλές φορές μένουν στην ίδια τη χώρα. Η Λάουρα ξέρει και τους αριθμούς. Πολλέ φορέ μπορεί να αρκεί να μετακινηθεί κανεί στο εσωτερικό λοιπόν τη ίδια τη χώρα, μπορεί να μην χρειαστεί να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παραμένοντα τουλάχιστον σε αυτή την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή τη χώρα του, μπορεί ο ακτιβιστή να έχει την ίδια ε, χρονική άτρακτο όπω οι συνάδελφοί του, να βρίσκεται δηλαδή στην ίδια ώρα με του συναδέλφου και αυτά που γράφει να πιάνουν τόπο. Είναι καλύτερο να μένει κανεί στην ίδια γεωγραφική ζώνη. Ξέρουμε, α πούμε, ότι ένα ακτιβιστή Κινέζο δεν μπορεί να παραμείνει στην ίδια γεωγραφική ζώνη ή στην περιοχή της Μεσογείου. Η Αίγυπτος έχει συνεργασία με όλες τις μυστικές υπηρεσίες όλων των σχετικών χωρών. Υπάρχουν ακτιβιστές που ε, συλλαμβάνονται στις χώρες του κόλπου μετά από παραγγελία της Αιγυπτιακής κυβέρνησης ας πούμε. Οπότε δεν χρησιμεύει πάντοτε αυτή η μετακίνηση, αλλά οι περισσότεροι από τους ακτιβιστές θέλουν να γυρνάνε πίσω στις χώρες τους. Πολλές φορές είναι η βασική επικεφαλής μιας ολόκληρης ομάδας ε, πληθυσμού ή κοινότητας. Οπότε δεν έχουν καμιά θέση στο εξωτερικό σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν ε, νέοι ηγέτες που αντικαθιστούν αυτούς που φύγαν ε, ως ακτιβιστές, ε, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη συσπήρωση στις περιπτώσεις αυτών των κοινοτήτων, των πληθυσμών. Πάντως είναι δύσκολο να φεύγει κανείς. Σπανίως μάλιστα υποβάλλουν τίμησεις ασύλου οι άνθρωποι αυτοί. Τώρα για τις απειλές αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε εσείς. Έχουμε καλέσει την κοινωνία των πολιτών ε, με όλα τα δίκτυα που υπάρχουν ε, να δούμε κατά πόσον μπορεί να υπάρξει ένα δίκτυο στα πλαίσια του rights and values, των δικαιωμάτων και αξιών. Κάτι που το χειρίζεται η Επιτροπή η δική σας, η Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη και μαζί νομίζω και η Γενική Διεύθυνση Just. Ω σήμερα ήταν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το δικαιώματα και αξίε για τη συνεργασία των διαφορετικών οργανώσεων των διαφορετικών χωρών, δεν θέματα πολιτισμού και παιδεία και το καθεξή. Βλέπουμε όμω στην Ευρώπη να έχουμε όλο ένα και περισσότερα προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, οπότε καλό θα ήταν να δημιουργηθεί ένα σχετικό μέτωπο. Διότι το κλασικό ευρωπαϊκό σχέδιο και πρόγραμμα για τη συνεργασία οργανισμών μεταξύ χωρών είναι πολύ ευέλικτο. Κάποιοι χρειάζονται έναν συνήγορο, κάποιο μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθεί, κάποιο μπορεί να χρειαστεί κάτι άλλο ακτιβιστή και πολύ, αμέ, πολύ ε, αμέσω. Πολύ γρήγορα. Εδώ λοιπόν μπορεί με αυτό το πρόγραμμα η παρέμβαση να είναι πολύτιμη όταν δεν γίνεται αλλιώ. Τώρα για τον κατάλογο των χωρών που αναφέρατε εσεί. Μίλησα για τέσσερι χώρε όπου υπάρχουν περισσότερε περισσότερες Ω προ τα ποσοστά είναι οι περισσότεροι θάνατοι αυτοί που καταγράφονται εκεί. Ε, υπάρχει βεβαίω πρόβλημα και με την Βενεζουέλα και την Ικαραγουά και πολλέ φορέ Λάουρα, έχουμε πρόβλημα και με τον αριθμό που αναφέρεται για τι χώρε αυτέ. Και πρέπει, με τα ποσά που έχουμε για τι χώρε αυτέ, να ε, έρθουμε να ζητήσουμε και συμπληρωματικά πολλέ φορέ. Ε, μπορεί σε μια περίοδο κρίση να έχουμε 152 αιτήσει ξαφνικά μαζεμένε. Γι' αυτό έχουμε αυτόν τον κατάλογο από κίνδυνων χωρών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν μπορούμε να τα στείλουμε και όλα εκεί, γιατί μετά δεν θα έχουμε για του υπόλοιπου. Θα ήταν καλό ίσω να βρίσκαμε μηχανισμού για να μπορούν να αυξηθούν τα ποσά σε περίπτωση κρίση, σε περίοδο κρίση, όπω αυτή που περιγράφω. Τώρα για τι θεωρήσει. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Θεωρήσεων ειδική εξαίρεση κατηγορία για τους ε, προασπιστές, τους ακτιβιστές. Αυτό που λέγεται ανθρωπιστική βίζα, κάτι είναι. Μια τρίμηνη ε, θεώρηση, σε τι διαφέρει από μια κλασική, μπορεί να εκδοθεί πολύ γρήγορα. Δεν είναι κλασική θεώρηση για την οποία χρειάζονται μήνες και μήνες. Πολλέ φορές ε, το πρόβλημα είναι ότι ακριβώ πρέπει να βγει ο άνθρωπος από τη χώρα κατευθείαν, αμέσως. Δεν υπάρχει διαδικασία όμω για του ακτιβιστέ, για την ειδική αυτή περίπτωση. Έχουμε να ασκήσει πολλές πιέσεις για να δημιουργηθεί μια τέτοια διαδικασία, αλλά υπάρχουν πολλές αντιστάσεις. Αντιστάσεις από τη Γενική Διεύθυνση Home. Ε, είπαμε επανειλημμένως, δεν είναι πάνω από 500-600 άτομα. Δεν θα ανοίξουμε την πόρτα σε ορδές μεταναστών που θέλουν να μπουν στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει πραγματικά κίνδυνος Τουλάχιστον προσπαθούμε να είμαστε σε συνεννόηση με χώρε που έχουν τέτοιου μηχανισμού για να πάρουμε το καλό παράδειγμα, αλλά στο ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Που να είναι και καλά ορισμένο και να μπορεί να λειτουργήσει και εύκολα. Να δώσω τώρα το λόγο, αλλά δεν απάντησα στην ερώτηση για τι απειλέ και τι μελλοντικέ προκλήσει. Θα δώσω το λόγο στην συνάδελφο. Η κυρία Μπατιστίνη έχει το λόγο. να συμπληρώσω λίγο τις πληροφορίες που σας έδωσε η συνάδελφος όσον αφορά την μετεγκατάσταση. Ένα από τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούμε είναι να διασφαλίσουμε ότι ο υπερασπιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορέσει να συνεχίσει την εργασία του. Όταν αξιολογούμε λοιπόν το αίτημα του, το αίτημα μετεγκατάστασης, αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο επιμένουμε. Πώ θα συνεχίσουν την εργασία του. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσει το έργο του. Αυτό δεν συμφέρει κανέναν. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε, αν θέλετε, έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μαζί του και η μετεγκατάσταση είναι ένα στάδιο μόνο της υποστήριξης που τους προσφέρουμε. Όπως σας είπα όμως είναι πιο πλήρης, πιο σφαιρική η υποστήριξή μας και ξέρετε ότι μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, έναν ηγέτη μια οργάνωση περάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκεται σε μια άλλη χώρα, βρίσκεται σε καθεστώ μετεγκατάσταση. Προσπαθούμε παράλληλα να βοηθήσουμε το έργο άλλων που εξακολουθούν επιτόπου και μπορούν να συνεχίσουν την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό και τον έφερε και η ΕΜΑ είναι ότι οι περασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσπαθούν να μετεγκατασταθούν σε τοπικό επίπεδο. Αν τους δοθεί δυνατότητα, προτιμούν να παραμείνουν στο εσωτερικό της χώρας, να πάνε σε μια γειτονική περιφέρεια, στην ίδια περιφέρεια. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να προωθήσουμε όλο και περισσότερο τοπικές πρωτοβουλίες παροχής καταφυγίων. Θεωρούμε ότι η μέθοδος αυτή είναι πολύ πιο αποτελεσματική και όντως ανταποκρίνεται στις ίδιες τις ανάγκες των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. και κατά αυτόν τον τρόπο, όπως σας είπα, μπορούν να συνεχίσουν το έργο τους. Και βέβαια η μετεγκατάσταση είναι μία ίστατη λύση. Προσπαθούμε μέσω άλλων λύσεων, μέσω άλλων μεθόδων, μέσω της κατάρτισης, μέσω κάποιων μέτρων ασφάλειας για τα εργαφεία τους, αλλά ακόμη και τις κατοικίες τους, να προσφέρουμε την προστασία αυτή προτού φτάσουμε στην ίστατη λύση που θα είναι η μετεγκατάσταση. Πολλές φορές όμως βλέπουμε ότι η μετακατάσταση είναι η μόνη ασφαλής διαθέσιμη λύση και γι' αυτό το λόγο και το όλο το ζήτημα της πολιτικής των θεωρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Ξέρετε ότι από το 2017, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ένα έγγραφο, μπορώ να σας το δώσω, στο οποίο περιλαμβάνονται κάποιες συστάσεις για το τι θα μπορούσαν να κάνουν τα κράτη-μέλη για να διευκολύνουν τη χορήγηση θεωρήσεων ε, όταν ε, δεν προβλέπεται καμία άλλη εναλλακτική, κανένα άλλο τρόπο πέρα από τη μετεγκατάσταση δηλαδή. Αναφερθήκατε επίσης και στις προκλήσεις. Καλύψαμε κάποιες από αυτές. Αλλά είπαμε ότι υπάρχουν και κάποιες νέες αναδυόμενες ε, προκλήσεις, όπως το να ποινικοποιούνται όλο και περισσότερο οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι καλούνται αυτή τη στιγμή να δραστηριοποιηθούν σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα εχθρικό, σε ένα περιβάλλον μιας ρητορικής που στρέφεται εναντίον τους, που τους παρουσιάζει σαν εχθρούς του κράτους ή τρομοκράτες. Καταλαβαίνετε ότι αν η κοινή γνώμη αρχίσει και τους προσεγγίζει, αρχίσει και τους αντιλαμβάνεται ως απειλή, τότε αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ το όλο έργο τους. Επομένω, αυτό θέλουμε να το καταπολεμήσουμε. Υπάρχουν επίση όλο και περισσότερε νομοθεσίε κατά τη τρομοκρατία υπέρ τη ασφάλεια που δυστυχώ προσπαθούν να δυσχεράουν και το ίδιο το έργο των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πολλέ φορέ αποτελούν τροχοπέδι ακόμα και για μα όταν προσπαθούμε να φτάσουμε του ανθρώπου αυτού και να του παράσχουμε βοήθεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί κατά την έγκριση νέων νομοθεσιών που ενδεχομένως να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και για να παρεμποδιστεί το έργο των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και βέβαια οποιαδήποτε αρνητική ρητορική εναντίον του θα πρέπει να σταματήσει. Τώρα όσον αφορά του μηχανισμού υποστήριξης, προφανώς χρειαζόμαστε κονδύλια, όχι μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Χρηματοδότηση η οποία θα διασφαλίσει ότι όντω μπορούν να επιτελούν το έργο τους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, και έχουμε εκπονήσει και το φυλάδιο αυτό το οποίο σας δείχνω, όπου δίνουμε και κάποιες συστάσεις σε εσά για το τι μπορεί να κάνετε ως βουλευτές για να μας υποστηρίξετε και εμάς και βέβαια να υποστηρίξετε τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ετέθη ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, δεν έχω διαθέσιμα όμως τα δεδομένα μαζί μου. Εμείς ως οι υπερασπιστέ των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουμε κάνει κάποια μελέτη η οποία να διασυνδέει την κατάστασή του με τα φαινόμενα διαφθορά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα που να κάνουν αυτό το συσχετισμό. Πάντω, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σα παρουσιάσω κάποια τέτοια δεδομένα. Ανάμεσα δηλαδή στην στάση τη κυβέρνηση και το βαθμό διαφθορά, μια κυβέρνηση ενό κράτου. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόσωπος Γενικής Διευθύνσης ΔΕΦΚΟ θέλει το λόγο. Α, με συγχωρείτε, ήθελα και εγώ να πάρω το λόγο, αν μου το επιτρέπετε, για να απαντήσω στο ερώτημα το οποίο απευθύνθηκε σε μένα. Προκειμένου να γίνει κανείς ένας δικηγόρος ειδικευμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα, τι μπορεί να κάνει. Πολύ καλή ερώτηση. Να σας δώσω την προσωπική μου εμπειρία. Το 2010 ήμουνα δικηγόρος ειδικευμένο σε εμπορικά ζητήματα και πραγματικά έβγαζα πολλά χρήματα τότε. Το 2010 όμως ε, αντιμετώπισα και εγώ και η οικογένειά μου τα δυσχερή αυτά γεγονότα που σας περιέγραψα και αποφάσισα να αλλάξω στη δεδρομία και να γίνω δικηγόρος υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα τελευταία 7 λοιπόν χρόνια δραστηριοποιούμε στον τομέα αυτό και είμαι πεπισμένος πια ότι ε, ακολούθησα το σωστό δρόμο ότι μπορώ πραγματικά μέσω της τροφής αυτής που έκανα στο επάγγελμά μου να έρθω σε επαφή με όλους αυτούς που σε τοπικό επίπεδο προσπαθούν να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να στραφούν κατά των συγκρούσεων και των διενέξεων. Πραγματικά αυτό οφείλει να κάνει κανείς. Τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να λειτουργήσουν στην πράξη μόνο όταν πραγματικά πιστεύουμε σε αυτά και τα υποστηρίζουμε στην Κυργυσία. Οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζονται πολλές φορές από το κράτος ως ξένοι πράκτορες. Πολύ συχνά έχω, έχω δεχτεί και εγώ επιθέσεις εξαιτίας των πελατών που έχω αναλάβει να υπερασπίσω. Νομίζω λοιπόν ότι αν είναι κανείς να γίνει δικηγόρος υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να οπλιστεί με υπομονή και θάρρος. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει, αν θέλετε, εδώ πέρα ε, ένα παγκόσμιο θεματολόγιο, προτεραιότητες οι οποίες να μπορούμε να τις προωθήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σημαντικότατο αυτό μήνυμα το οποίο στείλατε. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εν συνεχεία στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης προκειμένου να ολοκληρωθεί και η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Φαβιέτα Νέντε λέγομαι και είμαι αναπληρωτής τμήματάρχης ε, για τα θέματα αυτά στην DG Θα ήθελα επ' να ενημερώσω τα νέα μέλη της Επιτροπής σας για τους διάφορους μηχανισμούς χρηματοδότησης που έχουμε για αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, είναι παγκόσμιο το πεδίο. Κάποιος ρώτησε για κριτήρια. Είναι να είναι αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε τον ορισμό του ΟΗΕ που μπορεί να είναι άτομα, οργανώσεις που ενεργά προσπίζονται και υποστηρίζουν ειρηνικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τρεις τρόπους χρηματοδότησης. Έχουμε μια διευκόλυνση για την κρίση πρώτα απ' όλα, μια έκτακτη χρηματοδότηση που άμεσα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μικρές επιδοτήσεις για σύντομο χρόνο, ε, νομική συνδρομή, ιατρική ε, συνδρομή και άλλα τέτοια βράχη πρόθεσμα. Ε, περίπου 100 αγωνιστές ε, χρηματοδοτούμε από τη βάση αυτή και ε, μεταξύ αυτών μέλη οικογενειών και συγγενείς. Στη συνέχεια έχουμε το σύστημα προστασίας των αγωνιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το 2015, το Protect Defenders, δεν θα επεκταθώ, είναι πιο ε, ευρεία η στήριξη, δεν είναι κατεπίγουσα, έχουμε και μετακατάσταση εκεί και πολύ σημαντικό υποστηρίζουμε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ίδιες τις χώρες και προς στιγμή εργαζόμαστε πολύ σκληρά μαζί τους για να ανανεωθεί το πρόγραμμα για την επόμενη τριετία. Και τέλος, πολύ σημαντικό και αυτό, έχουμε τη διευκόλυνση ε, ανθρωπιστικών κρίσεων 3,5 εκατομμύρια ε, που είναι αναπερίπτωση και κατόπιν ετήσεως από κοινωνία των πολιτών ε, σε δύσκολες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει χώρος καν ή απειλείται. Και έχουμε και εμπιστευτικά έργα εκεί. Ήθελα να μιλήσω γιατί νομίζω ότι είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και το νέο μέσο που συζητούμε για τη συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να υπάρξει ένα χωριστό κονδύλι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Καταφέραμε να αυξήσουμε την πυρκοδότηση και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Αλλά θέλω να σα πω πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει αυτό ο μηχανισμό, ή αυτοί οι μηχανισμοί ε, ε, μακροπρόθεσμα, να είμαστε ευέλικτοι, να μπορούμε να λειτουργούμε και να ανταποκρινόμαστε στις μεγάλες και πολλές προκλήσεις που είναι καινούργιες και που ακούσατε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη του Κοινοβουλίου που είναι δεδομένη. Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τώρα. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι το σημείο σύνδεσμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του αγωνιστέ στην ΑΕΔ. Θα ήθελα να πω ότι η προστασία των αγωνιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει προτεραιότητα για την ΑΕΔ και με πολύ χαρά ακούω σήμερα ότι διάφορα από τα θέματα που ετέθησαν, όπω πώ μπορούμε να είμαστε πιο ενεργοί ε, σε θέματα περιβαλλοντικά ή στη διασπορά ε, ε, και αυτά είναι θέματα για μας, γι' αυτό θέλουμε να αναθεωρήσουμε τις ε, κατευθυντήριες γραμμές που είναι η βασική μας πολιτική για την υποστήριξη των ακτιβιστών μέσω των ειδικών μας αντιπροσωπιών και των πρεσβειών των, κρατικών, των κρατών μελών, αλλά έχουμε και ένα οδηγό για τις κατευθυντήριες γραμμές που το λέμε guidance note για το πώς μπορεί να υποστηρίζεται η διασπορά, να έχουμε περισσότερη ευαισθησία ως προς το φύλλο, ως προς τους αγωνιστές των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Τι γίνεται ε, με τους δικηγόρους. Ελπίζουμε να συνεργαστούμε όσο γίνεται. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Κάνουμε πολλά πράγματα και συζητούμε πολύ, δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά επίκειται μια εκδήλωση που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική γιατί πρέπει να συνεργαστούμε, είναι το Φόρουμ των ΜΚΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλες οι οργανώσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, συνεργαζόμαστε για να φέρουμε στις Βρυξέλλες αγωνιστές ε, για τα περιβαλλοντικά δικαιώματα για να συντονιστεί η δράση και να συνδεθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα με το περιβάλλον. Και ελπίζω και εκεί να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ε, και να προστατεύσουμε τους ε, ακτιβιστές αυτούς. Ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο στη Γιολάντα που ήθελε να μας μιλήσει για τη διαφθορά και την επιρροή που έχει αυτό ε, στους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατανοώ το εξής για τη διαφθορά. Στην περίπτωση του συζύγου μου, η διαφθορά προέρχεται άμεσα από την κυβέρνηση της πολιτείας. Για ποιο λόγο. Είναι συνένοχη με εκείνους που ε, αποψηλώνουν τα δάση μας. Γιατί το λέω αυτό. όταν υπάρχουν διάφορες ακροάσεις, δικαστικές διαδικασίες, είναι πολλές οι παρατυπίες. Ο Πάμπλο, ο άντρα μου, δεν θα έπρεπε να είναι φυλακή με βάση αυτή τη εντολή τη δικαστική. Αλλά επειδή η κυβέρνηση εποφελείται από εκείνου ε, και τα έχει κάνει πλακάκια ουσιαστικά που αποψηλώνουν τα δάση, πήγε στη δίκη και κάθε φορά που υπάρχει ακροαματική διαδικασία, κάθε φορά που έχει επισκεπτήριο στη φυλακή, ποιος έχει ε, το πάνω χέρι και την γνώση ειδοποιούν τους παραστρατιωτικούς και πηγαίνουν και αποκλείουν ε, ε, το δικαστήριο και αποκλείουν και τη, φυλακή και δεν αφήνουν κανένα να περάσει. Ούτε στην ακροματική διαδικασία, ούτε στο επισκεπτήριο. Διακόπτεται η ακροματική διαδικασία. Πώς είναι δυνατόν. Προφανώς είναι η κυβέρνηση της πολιτείας, αλλά και η μεξικανική κυβέρνηση κεντρική. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε ε, αυτό το θέμα και φυσικά ε, υπάρχει ζήτημα ε, σχέσης μεταξύ εξουσίας, διαφθοράς και αυτό επηρεάζει τους αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εδώ στην Υποπιτροπή μας σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη δουλειά σας, για το θάρρος σας ε, και για τη στράτευσή σας, αλλά και την ε, βούληση αυτή που έχετε να υποστηρίζετε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να περάσουμε στην κυκλισμένη των θύρων ε, συνεδρίαση με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης Βραζιλίας. Ευχαριστώ.